θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ένα σχέδιο έκθεσης για, το για την οποία θα δώσουμε το λόγο στην κυρία Κέλλερ που θα μας παρουσιάσει μια έκθεση ίδιας ε, πρωτοβουλίας που από την, ε, που προέρχεται από την Επιτροπή ΑΦΕΤ. Επειδή η μετανάστευση είναι πολύ σημαντικό θέμα για μας, Υπάρχουν τόσα θέματα που μπορούν να ανακύψουν από μία τέτοια έκθεση. Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, θα ήθελα να σε επενθυμίσω ότι η ΑΦΕΤ θα ψηφίσει στις 16 Μαρτίου, Φεβρουάριο 28 ψηφίζουμε εμείς και η προθεσμία υποβολής τροπολογιών είναι στις 2 Φεβρουαρίου στις 6 το απόγευμα. Γι' αυτό θα ακούσουμε καταρχήν τι έχει να μας πει η κυρία Κέλλερ. Thank you very much. Indeed, I would like to present... Θα ήθελα λοιπόν να σας παρουσιάσω το σχέδιο γνωμοδότησης και θα ήθελα να σας πω ότι η Επιτροπή ΑΦΕΤ συντάσσει μια έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας για τις μεταναστευτικές ροές ε, με ε, βάση την, ε, το μεταναστευτικά ρεύματα που προκύπτουν από την αστάθεια. Υπάρχει γνωμοδότηση ΔΕΒΕ και ΛΥΜΠΕ όπως βλέπετε από το έγγραφο. Αυτά τα δύο ε, αυτές οι δύο επιτροπές έχουν ασχοληθεί με την εξωτερική πτυχή της ε, μετανάστευσης. Και γι' αυτό εμείς θα θέλαμε να καλύψουμε την πτυχή της εργασίας. Δεν έχω εντάξει άλλες εξωτερικές ε, πτυχές. Αυτό μας ενδιαφέρει τι συμβαίνει στα σύνορα και αλλού. Θα δείτε τις ε, υποδείξεις μου στο έγγραφο. Προσπαθώ να κάνω συγκεκριμένες προτάσεις και προσπαθώ να είμαι όσο το δυνατόν πιο σαφής. Για παράδειγμα, ζητώ από την Επιτροπή να καταβάλει προσπάθεια στο θέμα της νόμιμης μετανάστευσης αναγνωρίζω ότι η Επιτροπή έχει κάνει πολλά, αλλά νομίζω θα πρέπει να ενδυναμώσουμε αυτή την πτυχή, διότι θα έχει επιπτώσεις και για το οργανωμένο έγκλημα. Στη συνέχεια υπάρχει μία παράγραφος για τη μετανάστευση που προέρχεται από τις κλιματικές αλλαγές εδώ χρειάζονται έρευνες, αλλά προτείνω να μας απασχολήσει το ζήτημα επικουρικής προστασίας για αυτούς τους μετανάστες, γιατί δεν έχουμε άλλους μηχανισμούς, δεν είναι πολιτικοί πρόσφυγες. Και γι' αυτό αυτή θα ήταν μια ενδιάμεση λύση πριν βρούμε μια μόνιμη ως, ε, για, ως προς τη σύσταση ενός συστήματος ελέγχου ενδιαφερόμαστε να δούμε κατά πόσο οι ετούντες άσυλο συμβαδίζουν με τον ε, κώδικα συνόρων Σέγγεν, να δούμε τι επιπτώσεις υπάρχουν γενικότερα και να δούμε και τις δραστηριότητες Frontex που σχετίζονται με τα μεταναστευτικά ρεύματα. Και υπάρχει και η μία σελίδα που είχαμε για το χρονοδιάγραμμα γνωμοδότησης. Αυτά είναι τα σημαντικότερα ζητήματα. Θα και ορισμένες άλλες τροπολογίες αλλά υπάρχει περιορισμός μίας σελίδας. Εάν εσείς βεβαίως θέλετε να υποβάλλετε τροπολογίες, μπορείτε να προβάλλετε πτυχές που δεν έλαβα υπόψη εγώ εδώ. Θα ήθελα όμως να σας πενθυμίσω ότι υπάρχει νέα προθεσμία η Δευτέρα Φεβρουαρίου, 2 Φεβρουαρίου, εξαιτίας των περιορισμών από πλευράς μετάφρασης. Είναι έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας Μιλάμε για τη μετανάστευση που προκύπτει από την αστάθεια. Θα ήθελα όμως να παραμείνουμε σε πτυχές που αφορούν την Επιτροπή μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδεις και την Γραμματεία για τη συνεισφορά της και παραμένω εδώ. Ευχαριστούμε κυρία Κέλλερ. Τώρα Αρχίζουν οι συζητή... Αρχίζει η συζήτηση, δεν ξέρω αν κάποιος θέλει το λόγο. Έχουμε κατάλογο. Ο κύριος Μισελ έχει το λόγο πρώτος. Κύριε Μισελ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι σε ένα τέτοιο θέμα, για ένα τέτοιο θέμα, θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι η ιστορία της ανθρωπότητας είναι η ιστορία των μεταναστευτικών ρεμάτων. Συμβαδίζουν. Δεν υπάρχει μεταναστευτική ροή μηδέν, μηδενική. Δεν υπήρξε ποτέ και δεν θα υπάρξει ποτέ. Νομίζω ότι αυτό είναι μια πρώτη κατάφαση γιατί πάντα τη βλέπουμε προβληματικά, δραματοποιούμε. Λέμε η μετανάστευση είναι πρόβλημα. Όχι, είναι ένα φυσικό είναι ένα φυσικό φαινόμενο και ως φιλελεύθερος θέλω να το τονίσω. Άρα δεν θα πρέπει να υπάρχει κανένα κατασταλτικό μέτρο που να προβληθεί. Δηλαδή οποιοδήποτε θέλει να μπορεί να δοκιμάσει αλλού την τύχη του. Γι' αυτό θα πρέπει να μπορεί με ευπρέπεια να μπορέσει να ασκήσει αυτό το δικαίωμά του. Γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να μας απασχολήσει κατά αυτό τον τρόπο η μετανάστευση. Όλοι μιλάμε για την κίνηση των πληθυσμών, είτε σαν χώρα διαμετακόμιση, είτε σαν χώρα υποδοχής. Σήμερα έχουμε 214 εκατομμύρια μετανάστευσα ανά τον κόσμο. Με την παγκοσμιοποίηση λοιπόν θα πρέπει να ξαναδούμε τις μεταναστευτικές ροές σε πιο αλληλέγγυα βάση έτσι ώστε όλα τα κράτη-μέλη να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν αυτή την πολιτική για να μπορούν όλοι οι άνθρωποι να ζουν με αξιοπρέπεια και ευπρέπεια. Θα πρέπει να έχουμε λοιπόν αυτή την προσέγγιση που να είναι πιο ευέλικτη. Δηλαδή να μιλάμε από πλευράς καθαρού κέρδους στις χώρες προέλευσης θα πρέπει να γίνουν περισσότερες επενδύσεις έτσι ώστε να δημιουργηθούν ε, θέσεις εργασίας, έτσι ώστε οι κάτοικοι να μην υποχρεωμένοι να μεταναστεύσουν. Να πρόκειται για μια προσωπική απόφαση, δηλαδή να αποφασίζει κανείς αν θέλει να μεταναστεύσει ή όχι. Υπάρχουν κέντρα διαχείρισης και πληροφόρηση των μεταναστών για να γνωρίζουν τις πραγματικές δυνατότητες νόμιμης μετανάστευσης και για να έχουν και τη σωστή κατάρτιση, ιδιαίτερα ως προς τη γλώσσα, και να καταπολεμήσουμε την παράνομη μετανάστευση, να προωθήσουμε τις μικροπιστώσεις για την έναρξη μιας οικονομικής δραστηριότητας. Η Γαλλία και η Ισπανία έχουν προβάλει ένα τέτοιο πρόγραμμα στο Μαλί. Και νομίζω ότι θα ήταν σκόπιμο να προωθήσουμε αυτή τη δομή ιδιαίτερα στις χώρες μετανάστευσης ή τις χώρες διαμετακόμισης για να μην, υπάρχουν, ε, να μην υπάρχει μια κατάσταση ρήξης και σύγκρουσης. Αυτό δεν το λέω επικριτικά, αλλά έχω την εντύπωση ότι πάντα όταν μιλάμε για τη μετανάστευση προσπαθούμε να δραματοποιήσουμε ένα ε, φαινόμενο το οποίο ε, είναι φυσικό. Δεν τυχαίο, δεν είναι δραματικό, δεν είναι προβληματικό, είναι ένα φυσικό φαινόμενο και θα ήθελα να σας πω ότι πολύ συχνά φαίνεται να υπονοούμε ότι ο μετανάστης δεν είναι το καλύτερο τμήμα ενός λαού. Δηλαδή ε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτοί που μεταναστεύουν είναι το καλύτερο μέρος ενός ε, πληθυσμού. Θέλουν να αναλάβουν την, ε, την ευθύνη των πράξεών τους και την τύχη στα χέρια τους. Αυτή είναι η βασική συλλογιστική. Δηλαδή η μετανάστευση είναι μια φυσική κατάσταση, ένα φυσικό φαινόμενο δεν αποτελεί εξορισμού πρόβλημα, Απλώ είναι, δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε εύκολα. Η κυρία Χολμάιερ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την ε, υποβολή του ε, κειμένου και χαίρομαι που έχουμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε και να ανταλλάξουμε απόψεις. Χαιρετίζω το ότι Όλες αυτές οι αιτίες για την ε, μετανάστευση αναφέρονται εδώ στο κείμενο ενδελεχώς. Εγώ θα ήθελα απλώς να ζητήσω να, για, την για το οργανωμένο έγκλημα να μην μιλούμε μόνο για το κατά πόσο υπάρχουν ε, νόμιμες δυνατότητες μετανάστευσης οι οποίες περιορίζουν την, ε, το οργανωμένο έγκλημα. Ας δούμε την το οργανωμένο έγκλημα και, αυτό, αυτό ασχολείται και η, ε, η, η, η άλλη επιτροπή του Κοινοβουλίου ε, για την ασφάλεια. Ας το δούμε και από άλλες πτυχές, γιατί ούτως ή άλλως μας απασχολεί συχνά. Είναι ένα σημαντικό σημείο, νομίζω, να μιλούμε και για τις ε, μεταναστευτικές ροές ε, που επηρεάζουν το οργανωμένο έγκλημα. Δεύτερον, θα ήθελα και σε σχέση με τους υπόλοιπους φακέλους που έχουμε για το συγκεκριμένο θέμα, να αναφέρω μία ανησυχία. Μερικές φορές ακούω κάποιες απόλυτες εκφράσεις για την διάσωση όλων αυτών των ανθρώπων που ε, διώκονται, κινδυνεύουν από κλιματικές αλλαγές ή ε, απειλούνται από κάτι. Ε, νομίζω ότι με αυτές τις απόλυτες εκφράσεις εδώ δεν θα μπορέσουμε να, λύσουμε, να σώσουμε τα τρία τέταρτα του πλανήτη. Νομίζω ότι αναλαμβάνουμε κάτι που η πραγματικότητα στο εσωτερικό των χωρών μας δείχνει ότι δεν γίνεται να γίνει. Πολλό δε μάλλον να γίνει και τα τρία τέταρτα του πλανήτη. Ας είμαστε υποδειγματικοί, ας είμαστε καλοί, αλλά πάλι ας μην είμαστε υπερβολικοί, ας μην θεωρούμε ότι, μπορούμε, ότι εμείς είμαστε σωτήρες όλου του κόσμου και ότι μπορούμε να λύσουμε ε, όλα τα προβλήματα όλου του κόσμου μόνο με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Um, Η λέξη αστάθεια με απασχόλησε ιδιαίτερα, ενώ πολλά θέματα δεν με βρίσκουν σύμφωνο σε αυτή την έκθεση δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπήρξαν ε, επιθετικοί πόλεμοι από την Δύση και ε, έμεσα στη Μέση Ανατολή δια πληρεξουσίου. Έπειτα υπάρχει ο παγκόσμιος καπιταλισμός που αντιμετωπίζει τους ανθρώπους σαν να ήταν μέσα παραγωγής, δηλαδή φτηνό εργατικό δυναμικό και ενθάρρυνση στις χώρες να ασχοληθούν με καλλιέργειες που αποδίδουν άμεσα παρά να έχουν μια μακρόπνοη πολιτική. Τώρα, κατά πόσο πρόκειται για μια ε, ε, πολιτική προς αποφυγή ή όχι, αυτό εξαρτάται από το εξής ε, βασικό ερώτημα. Οι διαφορετικοί άνθρωποι είναι, αποτελούν απότοκο διαφορετικών πολιτισμών. Άρα οι πολίτες του τρίτου κόσμου μπορούν να ε, κάνουν ουρά στα λιμάνια ή στα αεροδρόμια της Ευρώπης και μέσα σε μία γενιά να γίνουν Ευρωπαίοι, τότε όλα φαίνονται λογικά αν το δεχτείτε αυτό. Αν όμως βλέπετε διαφορετικούς πολιτισμούς, τρόπο ζωής, ως ε, απότοκο διαφορετικών λαών, τότε όταν εισάγεται το προϊόν αυτό του τρίτου κόσμου, δεν εισάγεται νέους Ευρωπαίους, αλλά φαίνεται το τρίτο κόσμο στα σύνορα της Ευρώπης και εντός Ευρώπης. Μούλτερ. Εντάχει. Πρόεδρε. Δεν ξέρω κατά πόσο κατανόησα καλά την κυρία Κέλλερ. Ίσως υπάρχουν διαφορετικές γνώμες για τα αίτια της μετανάστευσης. Αλλά μίλησε για τον μετανάστη, ε, ο οποίος γίνεται μετανάστης λόγω κλιματικών αλλαγών. Τι εννοεί όταν μιλάει για climate migrant. Η κυρία Έρνστ. Ευχαριστώ. Αυτό ακριβώς ήταν καλό γιατί η κυρία Κέλλερ ανέφερε και, τα, και τους πρόσφυγες. Γιατί αν δούμε τα κίνητρα για την ε, διαφυγή έχουν αλλάξει τα τελευταία χρόνια. Ας πούμε υπάρχουν πολλοί που ε, μετικούν λόγω, κλιματικών αλλαγών, λόγω έλλειψης νερού, λόγω απερίμωσης σε κάποιες περιφέρειες του κόσμου ή για μονοκαλλιέργειες ή λόγω μονοκαλλιεργειών που δεν μπορούν να εξασφαλίσουν πλέον την διατροφή. Υπάρχουν ε, πτυχές που έχουν ε, αλλάξει, έχουν εξελιχθεί τους τελευταίους αιώνες και κυρίως τις τελευταίες δεκαετίες. Και επίσης υπάρχουν ε, και νέες εξελίξεις στην όλη πολιτική προσφύγων και αυτές θα πρέπει να τις έχουμε υπόψη μας. Πρέπει καταρχάς αυτούς τους πρόσφυγες λόγω κλιματικών αλλαγών να τους δεχτούμε καταρχάς και αυτή την κατάσταση, αυτή δηλαδή την, αλλαγή των κλιματικών αλλαγών, το ότι αποτελούν ένα κίνητρο για αυτούς, ότι αποτελούν μια αιτία για ε, την ε, μετανάστευση, να, την, ε, να τη δεχτούμε. Και δεύτερον πρέπει να δούμε τι, γίνεται και με το ότι υπάρχουν ούτως ή άλλως ελλείψεις στι αναπτυξιακέ πολιτικέ παγκοσμίω για αυτού του ανθρώπου. Βεβαίω αυτό πρέπει να το δούμε και σε συνάρτηση με την μετανάστευσή τους. Έτσι ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους να ζουν στις χώρες που ζουν, όχι κάτω από βία, αλλά να προωθήσουμε δυνατότητες ανάπτυξης σε αυτές τις χώρες και για αυτούς τους ανθρώπους. Νομίζω ότι αυτά τα δύο θέματα θα πρέπει να τα σκεφτούμε. Ευχαριστώ. Thank you. Mrs. Fajon, got the floor. Yes, thank you very much. Κύριε ε, λυπάμαι που άργησα κάπως, γι' αυτό δεν παρακολούθησα την αρχή, αλλά θα πρέπει να μιλήσω ως κοιόδης. Είχαμε μια συζήτηση με τη Φραντσίσκα πολλές φορές και με άλλους συναδέλφους. Όπως είπε και ο προηγούμενος συνάδελφος, θα πρέπει να μας απασχολήσει η μεταναστευτική πολιτική. Και αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε ότι η αστάθεια είναι ευρύτατος όρος και δεν αρκεί να μιλάμε για κλίμα που οδηγεί το κλίμα, τις αλλαγές ε, του κλίματος που οδηγούν στη μετανάστευση, γιατί νομίζω ότι οι περισσότεροι μετανάστες προσέρχονται στην Ευρώπη λόγω οικονομικών και κοινωνικών συνθήκων. Γι' αυτό θα πρέπει να τονίσουμε περισσότερο τα μεταναστευτικά ρεύματα που απορρέουν από ολοκληρωτικά καθεστώτα, οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις φιλετικές διακρίσεις και να έχουμε μία πολιτική που να περιλαμβάνει όλες τις ε, πτυχές. Αυτό ακριβώς θα προβάλλω και εγώ γιατί νομίζω ότι η κυρία Κέλλερ έχει δίκιο Υπάρχουν και μετανάστες λόγω κλιματικών αλλαγών και στο μέλλον θα επιταθεί αυτό ακόμα περισσότερο. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι περισσότεροι μετανάστες προσέρχονται σήμερα στην Ευρώπη λόγω οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Αυτό θα ήθελα να τονιστεί. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω κανέναν άλλον να ζητάει το λόγο. Κυρία Κέλλερ, επανερχόμαστε σε εσά. Υποβλήθηκαν συγκεκριμένα ερωτήματα. Έχετε το λόγο για να απαντήσετε. Ευχαριστώ. Σύμφωνα με τον κύριο Μισελ, σε μεγάλο ποσοστό. Έχω ε, εδώ ότι θα πρέπει να πούμε ότι η μετανάστευση ήταν ένα διεθνές φαινόμενο που υπήρχε πάντοτε και που συνέβαλε και στην εξέλιξη της Ευρώπης και άλλων περιοχών. Και σημειώνω επίσης ότι είναι αδύνατο να σταματήσει κανένα τη μετανάστευση όπως είδαμε και με το Φρόνεξ όταν ήταν στις η νήσος. Οι μετανάστες πήγανε στη Μάλτα, όταν πήγανε το Frontex στη Μάλτα οι μετανάστες έρχονται μέσω της Ελλάδας Λοιπόν, θα πρέπει να μπορούμε να ελέγξουμε προ τα πού κινούνται και πώς, αλλά το να σταματήσουμε τελείως τη μετανάστευση είναι αδύνατο. <clears throat> Επίσης θα πρέπει να υπάρχει και μια θετική πτυχή ότι οι μετανάστες πολλές φορές ε, το βλέπουν σαν μια ευκαιρία. Το κάνουν εκούσια. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε και αυτό το στοιχείο. Θα προσπαθήσω να το βάλω στην ε, έκθεσή μου. Και επίσης τονίζω ότι οι περισσότεροι μετανάστες σε όλο τον κόσμο, οι περισσότεροι, δεν φτάνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι περισσότεροι πάνε είναι αλλού, στο Πακιστάν, στη Συρία, στις δικές τους περιφέρειες δηλαδή και περιοχές. Πολύ μικρός είναι ο που φτάνει εδώ στην Ευρώπη. Τα κέντρα ενημέρωσης είναι κάτι που ανέφερα πραγματικά στη συνάντηση ε, των σκιωδών. Ήταν θύματα του περιορισμένου χώρου που έχω για την έκθεση, αλλά θα μπορούσαμε να δούμε πώς θα το κάνουμε. Αν ε, θέλετε μπορείτε να υποβάλλετε συγκεκριμένες τροπολογίες. Ορισμός των μεταναστών κλίματος Είναι πολύ σαφές, νομίζω ο όρος. Είναι οι μετανάστες που αναγκάζουν να μεταναστεύσουν λόγω των επιπτώσεων του κλίματος της περιφέρειας τους. Ε, επίπεδο ε, ύδατος, ε, απερίμωση κλπ. Πολλές φορές η απερίμωση βέβαια δεν οφείλεται στην αλλαγή του κλίματος αλλά παραδείγματος χάρη στο ότι έχουν κόψει όλα τα δέντρα. Ε, Ε, τα Ηνωμένα Έθνα εκτιμούν ότι το 50% των εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων κινούνται ακριβώς λόγω κλιματολογικών αλλαγών και για άλλους περιβαλλοντικούς λόγους. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που παίζει σήμερα σημαντικό ρόλο στη μετανάστευση. Και οπωσδήποτε συνεχίσει. Προσπάθησα να αναφέρω τους κοινωνικονομικούς λόγους της μετανάστευσης. Δυστυχώς δεν είχα το χώρο που χρειαζόταν για να αναπτύξω το θέμα αυτό. Και επίσης άφησα επίδες κατά μέρος του τι μπορούμε να κάνουμε στις τρίτες χώρες για να άρουμε την ανάγκη μετανάστευσης για τους εκεί πολίτες. Γιατί εγώ προσπάθησα να δω τι μπορεί να γίνει στις ε, συνολικέ περιοχέ. Βέβαια, η ενσωμάτωση, οι διακρίσει είναι ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό για το οποίο δυστυχώ δεν υπήρχε καθόλου χώρο. Αυτά νομίζω λίγο πολύ. Και χαίρομαι να πάρω τις τροπολογίες σας 10 Φεβρουαρίου είναι η προθεσμία κατάθεση των τροπολογιών και περιμένω να ακούσω τις ιδέες σας. Ευχαριστώ κύριε Κέλλα, λέει Πρόεδρος. Δεν υπάρχουν άλλα σχόλια πάνω σε αυτό. Θα σας επιθυμήσουμε πάλι το χρονοδιάγραμμα. Θα ψηφίσουμε στις 28 Φεβρουαρίου και η προθεσμία για την αποβολή των απολογιών είναι 2 Φεβρουαρίου. 2 Φεβρουαρίου. Ωραία. Προχωρούμε στο επόμενο σημείο της μερικής διάταξης. Σημείο 9. Πλήρης εφαρμογή των διατάξεων και εκκλημένων του Σέγγεν στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. Έχουμε τον συνάδελφο Κάρλος Κοέλιο εισηγητή εδώ, αλλά θα ήθελα να σας υπενθυμίσω το τι έχει προηγηθεί. Με επιστολή του 12 Νοεμβρίου 2010 το Συμβούλιο μεταβίβασε με ένα σχέδιο απόφασης για την πλήρη εφαρμογή των ε, διατάξεων ΣΕΝΚΕΝ στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία μεταβίβασε λέω στις, ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για γνωμάτωση. Στις 16 Δεκεμβρίου η Νομική Επιτροπή ζήτησε από το Συμβούλιο να έχει πρόσβαση στην τελική αξιολόγηση και τι συστάσεις που γίνεται για κάθε χώρα, καθώς επίσης και πληροφορίες όσον αφορά πού βρίσκεται ο φάκελο αυτό τώρα για τις ε, συστάσεις προ την λόγω χώρε μέλη. Αυτά τα στοιχεία θεωρούνται απαραίτητα. Απαρά τα στοιχεία λέω για να ολοκληρωθεί η διαδικασία του των δυνατόν, πράγμα που επιθυμούμε. για να μπορέσει το Κοινοβούλιο να υιοθετήσει δική του γνωμοδότηση κατά τη διάρκεια τη Ολομέλεια του Φεβρουαρίου. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Κοέλιο, θα ήθελα να σα υπενθυμίσω ότι στο νέο προτινόμενο χρονοδιάγραμμα η εξέταση του σχεδίου της έκθεσης προεβλέπεται για τις 3 Φεβρουαρίου. 3 Φεβρουαρίου, επαναλαμβάνω. Και μετά μια σύνομη προθεσμία για τις τροπολογίες και η έγκριση της έκθεσης σε μια έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Λίμπε στις 14 Φεβρουαρίου στο Στρασβούργο. Τώρα θα ακούσουμε τον εισηγητή μας, τον κύριο Κοέλιο και μετά θα συζητήσουμε το θέμα. Και θα ακούσουμε επίση απόψει των εκπροσώπων τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και του Συμβούλιο που είναι παρόν εδώ. Παρακαλώ, κύριε Κοέλιο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη από τους ε, συναδέλφους, διότι δεν θα είμαι τόσο διπλωματικός και θα είμαι απόλυτα σαφής ως προς αυτά που θέλω να πω θα πρέπει να μιλήσω για το σεβασμό προς το Κοινοβούλιο. Δεύτερον, το τι συμβαίνει, ποια είναι τα τεκτενόμενα και τι πρέπει να κάνουμε. Ως προς το σεβασμό του Κοινοβουλίου. Θα αρχίσω από αυτό που μόλις πενθύμησε ο Πρόεδρος. Το Συμβούλιο ζήτησε να ακούσει την απόψή μας το Νοέμβριο, το Δεκέμβριο. Εγώ διορίστηκα εισηγητής και στις 16 Δεκεμβρίου ζητήσαμε τα έγγραφα, για να είμαστε απόλυτα σαφείς. Εμείς είχαμε την πολιτική θέληση ώστε η Βουλγαρία και η Ρουμανία να μπουν στο χώρο Σέγγεν. Αυτή είναι και η φιλοδοξία των δύο αυτών χωρών από τη στιγμή που έγιναν πλήρη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως, για να φτάσουν να ενταχθούν στο χώρο Σέγγεν θα πρέπει να ελεγχθούν όροι ασφάλειας και συνθήκες ασφάλειας. Σύμφωνα με τους ισχύοντες ε, κανόνες δεν μπορούμε να κάνουμε αυτή την ε, αξιολόγηση. Υπεύθυνε μία εβδομάδα που εξαρτάται από το Συμβούλιο. Αυτά τα έγγραφα θα πρέπει να επιδοθούν στο Κοινοβούλιο. Εμείς δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε την θετική ή αρνητική έκβαση της αξιολόγησης αν δεν έχουμε πρόσβαση στα έγγραφα αξιολόγησης. Στις 16 Δεκεμβρίου ζητήσαμε αυτά τα έγγραφα από το Συμβούλιο. Σήμερα βρισκόμαστε στην 25η Ιανουαρίου και δεν έχουμε ακόμα απάντηση από το Συμβούλιο. Δεν έχουμε λάβει απάντηση από το Συμβούλιο από τις ε, άτυπες οδούς μάθαμε ότι το Συμβούλιο βρίσκεται στην απαρχή μιας απάντησης, η οποία λέει ότι τα έγγραφα αυτά δεν θα δοθούν στο Κοινοβούλιο. Θα είναι διαθέσιμα σε μια κλειστή αίθουσα του Συμβουλίου. Και αν θέλουμε εμείς μπορούμε να μεταβούμε στο Συμβούλιο για να ελέγξουμε αυτά τα έγγραφα. Αυτό σημαίνει ο πρόεδρος της Επιτροπής οι συντονιστές πολιτικών ομάδων και ο εισήγητης ούτε καν οι δεν έχουν άδεια να συμβουλευτούν αυτά τα έγγραφα στο Συμβούλιο. Και κανένα από τα μέλη αυτά, αυτής της Επιτροπής, το μέλη που θα πρέπει να ψηφίσουν, δεν θα είναι σε θέση να, δεν θα είναι σε θέση να γνωρίσουν τα έγγραφα έτσι ώστε να αξιολογήσουμε εάν πληρούνται οι όροι ασφάλειας για την προσχώρηση. Αυτό το θεωρώ απαράδεκτο, Πρόεδρε. Το θεωρώ απαράδεκτο. Δεν είναι προσωπικό το πρόβλημά μου. Γιατί εγώ έχω πρόσβαση στο, στα έγγραφα. Το πρόβλημα είναι του Κοινοβουλίου. Δηλαδή αυτό που είναι δικό μου πρόβλημα είναι και δικό σας και αφορά και τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως πρόεδρο αυτού του σώματος. Υπάρχει ένα θέμα ρύθμισης σχέσεων μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Έμαθα ότι ο πρέσβης της ε, ε, Ρουμανίας, επειδή δεν είναι ικανοποιημένος ε, από αυτή την κατάσταση, θα ζητήσει να μην έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα τα έγγραφα, δηλαδή να μειώσει αυτό το κλιμάκιο για να μην βρισκόμαστε σε αυτή τη δύσκολη θέση. Τα πράγματα δεν είναι καθόλου σοβαρά τη στιγμή που ο πρέσβης μιας χώρας ζητά να μειωθεί ή να αφαιρεθεί ο εμπιστευτικός χαρακτήρας από τα έγγραφα επειδή δεν είναι ε, αγαστές οι σχέσεις μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Θα έπρεπε να μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε αυτά τα έγγραφα. Η Κομισιόν μας είπε με email ότι τα έγγραφα που έχει εκείνη θα ε, διατεθούν στο Κοινοβούλιο. Ε, χαίρομαι γιατί ο ανώτερος αξιωματούχος της Επιτροπής το κατάφερε αυτό, αλλά τα έγγραφα αυτά δεν είναι το σύνολο των εγγράφων για την αποτίμηση της κατάστασης και τα έγγραφα αυτά δεν έχουν ακόμα ψηφιστεί. Ίσως δεν αποτελούν δηλαδή τελική έκδοση και δεν ξέρουμε κατά πόσο θα εγκριθούν στις 28 Ιανουαρίου. Αλλά τίποτα δεν μας εγγυάται ότι τα έγγραφα αυτά που έφτασαν από την κυρία Καπιτάνη, από την Κομισιόν, δεν ξέρουμε κατά πόσο αυτά θα είναι τα έγγραφα που θα εγκριθούν τελικά από το Συμβούλιο. Αυτό είναι και το πρώτο θέμα. Δεν ε, σέβεται το Συμβούλιο το Κοινοβούλιο. Δεύτερον, επί του περιεχομένου τώρα και σύμφωνα με τις πληροφορίες που προήλθαν ατύπως, βλέπουμε ότι δεν θα υπάρχουν προβλήματα με τη Ρουμανία. Υπήρχαν προβλήματα σε επίπεδο Σέγγεν με ορισμένες προειδοποιήσεις που σχετίζονται με το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Αυτά τα θέματα ε, έχουν επιληθεί από ό,τι φαίνεται, προφανώς αν δεν είναι σίγουρο. Υπάρχουν όμως προβλήματα με τη Βουλγαρία, ιδιαίτερα ως προς τον έλεγχο τον επίγειο έλεγχο μεταξύ Βουλγαρίας και Τουρκίας. Ίσως οι Βούλγαροι αντιμετωπίζουν πραγματικό πρόβλημα, είπαν θα το επιλύσουν τάχιστα. Ε, στο μεταξύ οι δύο υπουργοί, ο Γερμανός και ο Γάλλος, υπέβαλαν μία επιστολή λέγοντας ότι υφίστανται ορισμένα προβλήματα ως προς την καταπολέμηση της διαφθοράς που θα μπορούσαν να προδικάσουν την αίσια έκβαση αυτού του θέματος. Θα ήθελα να είμαστε απόλυτα σαφείς ως προς το πρόβλημα του Συμβουλίου. Αν οι Υπουργοί θέλουν να το αναβάλουν, όχι αυτό δεν είναι δικό μας πρόβλημα. Το δικό μας πρόβλημα είναι ότι πρέπει να γνωμοδοτήσουμε επί μιας πρωτοβουλίας. Δηλαδή να προσχωρήσουν στο χώρο Σέγγεν αυτές οι δύο χώρες. Γι' αυτό εμείς θα πρέπει να γνωμοδοτήσουμε γνωρίζοντας όλα τα στοιχεία του φακέλου. Τρίτον και τελευταίο. Τι είναι, τι θα κάνουμε. Τι με λιγενέστε. Κατά την άποψή μου θα πρέπει να μεταβούμε στο ανώτερο επίπεδο και να ζητήσουμε πρόσβαση στα έγγραφα. Αυτό είναι σημείο εκκίνησης κατά την άποψή μου και τι μπορεί να συμβεί. Ένα από τα δύο μπορούν να συμβούν. Η πρώτη κατάσταση είναι να μην λάβουμε τα έγγραφα στο εγγύς μέλλον και το Συμβούλιο που αντιμετωπίζει προβλήματα λήψης απόφασης, γιατί σας υπενθυμίζω ότι το Συμβούλιο πρέπει να αποφανθεί ομόφωνα και μόνο ομόφωνα, το Συμβούλιο θα μπορούσε να μας πει ότι ότι το πρόβλημα που ε, αντιμετωπίστηκε είναι ίσονος σημασίας, διότι το Συμβούλιο δεν μπορεί να λάβει καμία απόφαση αν δεν αποφανθεί, αποφανθεί το Κοινοβούλιο. Άρα η καθυστέρηση του Κοινοβουλίου θα ήταν δικαιολογία για το Συμβούλιο. Άρα θα είμαστε αναγκασμένοι να αποδιώξουμε το θέμα από το Κοινοβούλιο αν δεν μπορούμε να προβούμε σε μία αποτίμηση ουσίας, δηλαδή αν δεν έχουμε τα έγγραφα του Συμβουλίου. Και θα σας πρότεινα να γνωμοδοτήσουμε λέγοντας ότι δεν μπορούμε να γνωμοδοτήσουμε. Δηλαδή, να εγκρίνουμε γνωμοδότηση λέγοντας ότι εφόσον δεν είχαμε πρόσβαση στα έγγραφα για να γνωμοδοτήσουμε επί της ουσίας, δεν θα γνωμοδοτήσουμε. Άρα επίσημα γνωμοδοτούμε, γνωμοδοτούμε ότι δεν γνωμοδοτούμε, άρα γνωμοδοτούμε, κατά την αριστοτέλεια λογική, και νομίζω ότι έτσι μπορούμε να ξεφύγουμε από το πρόβλημα, δηλαδή αυτό το πρόσκαμα το, πρόσκαμα το καθαρά διοικητικό, το αντιπαρερχόμαστε. Αν έχουμε τώρα τις ε, εκθέσεις, τότε υπάρχουν τρία ενδεχόμενα. Η έκθεση θα αναφέρει ότι τα δύο κράτη-μέλη μπορούν να προσχωρήσουν στο χώρο Σέγγεν. Τότε εμεί θα συμβαδίσουμε. Ή η έκθεση θα πει ότι καμία από τις δύο χώρες δεν είναι σε θέση να προσχωρήσει τότε θα πρέπει να προβούμε σε μια πολιτική αξιολόγηση για το πώς ερμηνεύουμε αυτές τις εκθέσεις, αυτή την έκθεση. Και θα δούμε κατά πόσο έχουν αλλάξει τα δεδομένα, δηλαδή έχουν ε, ανταποκριθεί οι χώρες για την άρση των δυσχεριών ή θα πρέπει να γνωμοδοτήσουμε ότι υφίσταται ακόμα αυτή η κατάσταση, γι' αυτό καμία χώρα δεν μπορεί να προσχωρήσει το χώρο Σέγγεν. Υπάρχει όμως και μια τρίτη πιθανότητα ότι δηλαδή μία χώρα πληρεί τους όρους και η άλλη όχι. Εάν επαληθευτεί αυτή η κατάσταση, εμείς θα πρέπει να προβούμε σε μία χρονική αξιολόγηση. Δηλαδή να κατανοήσουμε κατά πόσο πρόκειται για μία κατάσταση που θα παραταθεί μέσα στο χρόνο ή μπορεί να επιληθεί σύντομα. Εάν ναι, τότε θα ήταν σκόπιμο να προσχωρήσουν και οι δύο χώρες. Εάν όμως παραταθεί το θέμα, τότε θα πρέπει να δούμε κατά πόσο η χώρα που πληρεί τους όρους μπορεί να προσχωρήσει χωρίς να υπάρξουν δυσκολίες για τη δεύτερη χώρα και χωρίς τα σύνορα μεταξύ των δύο χωρών να πληρούν τις παραμέτρους ασφαλείας όπως προαπαιτεί ο χώρο Σέγγεν. Ζήτω συγγνώμη, δεν ήμουν καθόλου διπλωματικό στην παρέμβασή μου, αλλά σας έδωσα όλα τα στοιχεία εκτίμησης. Θα πρέπει να υπάρχει σεβασμός προς το Κοινοβούλιο, να δούμε τι γίνεται με τις διμερείς μας σχέσεις με το Συμβούλιο και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε επί της ουσίας. Έτσι έχει η κατάσταση επί του θέματος. Σας ευχαριστώ. Thanks εγώ ευχαριστώ κύριε Κοέγιο για τις εξηγήσεις σας και τη θέση που έχετε σε αυτή την ε, γνωμοδότηση. Να σας θυμίσω απλώς ότι εγώ ως πρόεδρος έχω τονίσει τη σημασία αυτού που είπατε το να υπάρχει δηλαδή πλήρης πρόσβαση σε όλα τα σχετικά έγγραφα που σχετίζονται με την απόφαση που πρέπει να ληφθεί για, την, για το κατά πόσο πληρούνται οι προϋποθέσεις για το κεκτημένο Σέγγεν και για την Βουλγαρία και για την Ρουμανία. Σε κάθε παρέμβαση, σε κάθε ομιλία που έχω κάνει, και σε κάθε συζήτηση που έχω κάνει με όλους τους εκπροσώπους και από την Κομισιόν και από το Συμβούλιο και επί τη ευκαιρία της παρουσίασης του προγράμματος της Ουγγρικής Προεδρίας και με τον μόνιμο αντιπρόσωπο, τον πρέσβη της, Ουγγαρίας και τη δική του ομάδα και επί τη ευκαιρία του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών που έγινε στη Βουδαπέστη το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Το είπα και το ξαναείπα. Είναι λοιπόν θέμα αρχής. Δεν είναι το κατά πόσο είναι δίκαιο το αίτημα ή όχι, είναι θέμα αρχής. Είναι θέμα του ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι η Λισαβόνα ισχύει, ότι το Κοινοβούλιο έχει λόγο, ότι μπορεί να παίξει αποφασιστικό ρόλο και ότι πρέπει να έχει πλήρη πρόσβαση σε όλα τα σχετικά έγγραφα για να μπορέσουμε και εμείς να λάβουμε απόφαση. Πλήρη πρόσβαση <clears throat> λοιπόν. Όχι ιονή πρόσβαση σε κάποια επιλεγμένα μέλη της Επιτροπής, πλήρη πρόσβαση σε όλα τα μέλη. Για να μπορούμε να λάβουμε σωστές αποφάσεις. Και να προσθέσω επίσης ότι κάθε επιστολή που έχει στελεί από την Γραμματεία και κάθε βήμα που έχει γίνει από την Γραμματεία της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ έχει γίνει εν γνώση του Προέδρου της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Γιατί ξέρουμε ότι είναι ακριβώς θέμα αρχής αυτό το οποίο συζητούμε εδώ. Μιλούμε για την ε, αγαστή συνεργασία. Τα θεσμικά όργανα πρέπει να επικουρούν το ένα το άλλο. Το Συμβούλιο λοιπόν και το Κοινοβούλιο, οι δύο φορείς νομοθετικού έργου στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επικουρούν ο ένας τον άλλον. Λοιπόν, ε, τούτου δίνω το λόγο σε όποιον τον θέλει για να μιλήσει και μετά θα ακούσουμε από την Προεδρία και από την Κομισιόν. Πρώτα η κυρία Βέμπερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ που τόσο ενεργά έχετε λάβει το ρόλο του Προέδρου και προσπαθείτε ώστε οι, τα μέλη της Επιτροπής να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Γιατί από ό,τι φαίνεται στο Συμβούλιο και αν ε, το λέει ο κύριος Κοέγιο ε, δεν το, αν λέει ότι δεν μίλησε πολύ διπλωματικά δεν, περιμένετε να δείτε τι θα πω εγώ το Συμβούλιο αυτό που κάνει είναι να προσπαθεί να παρεμποδίσει το ρόλο του Κοινοβουλίου τον οποίο ορίζει η συνθήκη ανεξάρτητα από το γεγονός ότι είμαστε σε συναπόφαση ή αν είναι γνωμοδότηση αυτή που πρέπει να δώσουμε εμείς στο Συμβούλιο, η δική μας δουλειά είναι να εργαστούμε επί αυτών των εκθέσεων. Αυτή τη στιγμή στο Συμβούλιο έρχεται με δρακόντια μέτρα και δεν μας επιτρέπει να έχουμε πρόσβαση σε έγγραφα, αυτό σημαίνει ότι δεν θέλει να μας αφήσει να κάνουμε τη δουλειά μας. Εκτός εάν το Συμβούλιο θεωρεί ότι εμείς εδώ ερχόμαστε για να κάνουμε τα ψώνια μας, να πιούμε καφέ και να δούμε τους φίλους μας. Όχι. Είμαστε σε ένα κοινοβούλιο και τρέχουμε από τη μία αίθουσα στην άλλη, από τη μία συνεδρία στην άλλη και προσπαθούμε να ανταποκριθούμε στα καθήκοντά μας. Πρέπει να πω όμως ότι είναι η πρώτη φορά που βρισκόμαστε σε μια τέτοια κατάσταση. Έχουμε χρονοδιάγραμμα και δουλεύουμε με σενάρια. Τι θα γίνει αν. Ε, είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Δεν είναι απλώς απαράδεκτο είναι απίσταυτο, ε, είναι, ξεπερνάει την όποια φαντασία. Δηλαδή το Συμβούλιο τι ακριβώς θεωρεί ότι, πρέπει ότι κάνουμε εμείς εδώ. Μέχρι πριν από λίγες ημέρες εγώ έκανα ό,τι μπορούσα για να Πιστώ ότι αυτή ήταν έτσι μια κατάσταση που δεν σχετίζεται με το συγκεκριμένο φάκελο. Είναι ένα θέμα ισχύω μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Το Συμβούλιο δεν καταλαβαίνει ότι είμαστε, έχουμε ίση αξία Κοινοβούλιο και Συμβούλιο πια. Αλλά πρέπει να πω ότι έχοντας δει και σε πολιτικό επίπεδο τις επιστολές που ανταλλάγησαν, με το Συμβούλιο, ε, και ό,τι έγινε, νομίζω ότι θα αρχίσω κι εγώ να πιστεύω τις θεωρίες συνωμοσία. Δηλαδή, το Συμβούλιο προσπαθεί να μας εμποδίσει ε, να έχουμε πρόσβαση σε, αυτή την, ε, σε αυτές τις πληροφορίες ένα τμήμα μιας γενικότερης συνωμοσία για να μην δώσει θετική γνώμη το Κοινοβούλιο. τι να σας πω, αναρωτήθηκα κάποια στιγμή. Νομίζω ότι αυτό το θέμα πρέπει να το λύσουμε σε επίπεδο θεσμικό. Αύριο στους συντονιστές εγώ θα καταθέσω επίσημο αίτημα να, ζητήσουμε από τον, επίδροπο, από τον πρόεδρο συγγνώμη, Μπούζεκ να στείλει επιστολή στην, στον πρόεδρο της Κομισιόν στο, συμβουλίο, στο πρόεδρο του Συμβουλίου συγγνώμη, και να ζητήσει να αφήσουμε το Κοινοβούλιο να κάνει τη δουλειά του. Είναι απαράδεκτο αυτή τη στιγμή δύο ε, οι υψηλοί αξιωματούχοι του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου ασχολούνται με αυτό το θέμα και εγώ, μια εκλεγμένη βουλευτής από το λαό της Ευρώπης, πρέπει να υποκύψω στις επιθυμίες ενός δημοσίου υπαλλήλου του Συμβουλίου. Συγγνώμη, αυτό πρέπει να το λύσουμε. Γι' αυτό θα πρέπει ο πρόεδρος Μπούζικ να στείλει επιστολή στο Συμβούλιο και στην Προεδρία την Ουγγρική και η Προεδρία θα πρέπει να δώσει την απάντηση στο πρόβλημα αυτό τι θα κάνουμε με τους φακέλους αυτούς, ιδέα δεν έχω. Εγώ μάλιστα είμαι και σκιώδης εισηγήτρια, οπότε δεν έχω ούτως ή άλλως πρόσβαση. Αλλά ως συντονίστρια έχω πρόσβαση. Αλλά οι συνάδελφοί μου τι θα κάνουνε. Που θέλουν να έρθουν να ψηφίσουν για την έκθεση αυτή. Δηλαδή τι γίνεται σε αυτό το, ποιοι είμαστε εμείς σε αυτό το κοινοβούλιο, έχουμε αλλάξει τελείως τους κανόνες του παιχνιδιού. Νομίζω ότι πρέπει να το λύσουμε το θέμα αυτό, άπαξ και διαπαντός. Αυτά προς το παρόν. Και βεβαίω θα συνεργαστώ πολύ στενά με τον κύριο Κοέγιο για την έκθεση αυτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ως ε, σκιώδης από πλευράς ε, σοσιαλιστών και δημοκρατών θα ήθελα να πω και εγώ να κάνω κι εγώ ορισμένα σχόλια. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Κοέλιου για την σαφή ανάλυση σε σχέση με την κατάσταση μέχρι τώρα όπως αποτίμησε δηλαδή τη συνολική κατάσταση. Θα ήθελα ο κύριος Κοέλιου να προβλέψει σύντομα μία συνεδρίαση με τους σκιώδεις έτσι ώστε να εκπονήσουμε μία κοινή στρατηγική ανεξάρτητα από την πολιτική ομάδα στην οποία ανήκουμε. Εμείς που έχουμε εκλεγεί άμεσα θα πρέπει να απαιτήσουμε το σεβασμό προς εμάς. Για τους Βούλγαρους και τους Ρουμάνους δεν πρόκειται απλώς για μία επιθυμία, πρόκειται για νομική επιταγή, όπως είπε και ο κύριος Κοέλιου, όπως προβλέπει και η συνθήκη της Λισαβόνας. Και βεβαίως θα πρέπει να αποφανθεί ομόφωνα το Συμβούλιο μετά από αποτίμηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μετά από τις συστάσεις της ομάδας που έχει συσταθεί στο Συμβούλιο. Από τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι τώρα, από τις άτυπες πληροφορίες, φαίνεται ότι η Ρουμανία πληρεί όλους τους όρους, ενώ η Βουλγαρία αντιμετωπίζει προβλήματα παρά το γεγονός ότι το Συμβούλιο δεν μας διέθεσε τις εκθέσεις αξιολόγησης, θεωρούμε ότι μπορούμε να ε, δράσουμε, να αναλάβουμε μία δράση, να πιέσουμε το Συμβούλιο έτσι ώστε να μας δώσει τα έγγραφα αυτά. Πιστεύουμε λοιπόν ότι αυτή θα πρέπει να είναι η επίσημη θέση μας. Βεβαίως γνωρίζουμε την επιστολή της γαλλικής κυβέρνησης μαζί με τη γερμανική και έγινε λόγος για ε, μια επικίνδυνη κατάσταση στα σύνορα Βουλγαρίας με την Τουρκία. Και ελέγχθη ακριβώς ότι γι' αυτό δεν μπορεί να προσχωρήσει η Βουλγαρία στο Σέγγεν. Αλλά εμείς έχουμε πρόσβαση στα στοιχεία του συστήματος Σέγγεν από πέρσι. Δηλαδή πληρούμε τους όρους και τις προδιαγραφές. Νομίζω λοιπόν ότι η ρουμανική κυβέρνηση έχει επαληθεύσει την κατάσταση και ξέρετε ότι γνωρίζουμε και εσωτερικούς κλειδονισμούς εξαιτίας της ε, ε μιας κατάστασης κοινωνικών αναταραχών στη Ρουμανία. Εν πάση περιπτώσει αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να ενσωματωθούμε στο χώρο του Σέγγεν. Όλα αυτά τα στοιχεία επαληθεύτηκαν από το Συμβούλιο οι αποτιμήσεις και οι αξιολογήσεις ήταν σωστές. Όλες οι άλλες αιτιάσεις δεν είναι σωστές. Και νομίζω ότι οι αντιρρήσεις της Γερμανίας και της Γαλλίας σχετίζονται με την αντίθεσή τους προς τη ρουμανική κυβέρνηση και δεν σχετίζονται με αντιρρήσεις επί της ουσίας. Δεν νομίζω λοιπόν ότι μπορούν να προβληθούν τέτοιες αντιρρήσεις. Αυτό εντάσσεται στις ε, διμερείς σχέσεις και αφορά και το θέμα αντιμετώπισης των Ρωμά. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να τους υποστηρίξουμε όπως ορίζει το ευρωπαϊκό δίκαιο. Εν πάση περιπτώσει, το ευρωπαϊκό Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να βασιστεί στα συμπεράσματα των αξιολογήσεων του Συμβουλίου. Γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να μας δοθεί άμεση πρόσβαση σε αυτές τις εκθέσεις. Αυτή είναι η καλύτερη λύση και θα πρέπει να βασιστούμε σε αντικειμενικά στοιχεία αποκλειστικά και τίποτα άλλο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Έντσου. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Κοέλιου για την έκθεσή του. Νομίζω ήταν ιδιαίτερα διπλωματικός. Δεν μπορεί να μην έχουμε την δυνατότητα να έχουμε πρόσβαση σε αυτά τα έγγραφα και να μην ξέρουμε επί τίνος ψηφίζουμε. Το θέμα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο σε σχέση με την προσχώρηση της Ουγγαρίας στον χώρο Σέγγεν την διαδικασία την παρακολούθησα εκ του και είδα ότι είχε μεγαλύτερη επίπτωση στον πληθυσμό από την ίδια την προσχώρηση της χώρας μου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι έτσι ο κόσμος έβλεπε ε, εν της πράγμαση τι αλλαγές έχουν επέλθει και πώς διευκολύνεται η καθημερινή του ζωή. Και εάν υπάρχει ίση μεταχείριση θα πρέπει να είναι ίση ως προς όλες τις πτυχές. Έχει μεγάλη σημασία για, τον, για τους λαούς αυτών των χωρών γιατί οι, οι λαοί αυτοί υποστηρίζουν την προσχώρηση στο χώρο Σέγγεν. Άρα ο ρουμανικός και βουλγαρικός λαός θα πρέπει να μπορούν να προσχωρήσουν στο χώρο Σέγγεν και θα πρέπει ο πρόεδρος Μπούζεκ να λάβει θέση ως προς τη στάση του Συμβουλίου και να ζητήσει να έχουμε άμεση πρόσβαση σε αυτά τα έγγραφα για να μην επιδεινωθεί η παρούσα κατάσταση. Σόμερ. Σόμερ. Yes. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte mich... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και εγώ τον συνάδελφο Κοέλιο. Ε, δεν μπορούμε να είμαστε διπλωμάτε. Ε, άλλωστε δεν είμαστε διπλωμάτε. Πολιτικοί είμαστε. Πρέπει να λέμε την άποψή μα. Ξέρω ότι εσεί γενικώ έχετε έτσι, μια παράδοση ε, στον τρόπο που εκφράζεστε στη χώρα σα, αλλά από εκεί που έρχομαι εγώ, εντάξει, μπορούμε να είμαστε και λίγο πιο θρασεί. Αλλά πρέπει να συζητήσουμε το θέμα αυτό. Στην πολιτική πρέπει να ακούγονται οι απόψει. Λοιπόν, είναι πραγματικά ξεδιαντροπιά αυτό που συμβαίνει. Να μην έχουμε την, ε, τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε. Ή να δίνονται απλώς, να δίνεται πρόσταση, πρόσβαση σε κάποιους, σε ένα και στο δωμάτιο, σε λίγους επιλεγμένους. Και μάλιστα και στο Συμβούλιο μόνο. Δηλαδή πρέπει και να πάμε κιόλα. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε και εδώ. Έχει ξαναγίνει. Εγώ είναι η τρίτη μου θητεία τα πρώτα δέκα χρόνια μόνο νομοθετική δουλειά έκανα, οπότε ξέρω τι σημαίνει. Αυτό λοιπόν το παιχνιδάκι με το Συμβούλιο το γνωρίζω, αλλά αυτό που γίνεται τώρα και με την ε, ε, συνθήκη της Λισαβόνας, ε, που έχουμε μέσω αυτής την συναπόφαση εδώ η ΛΥΜΠΕ, δεν, το, δεν το έχω ξαναδεί, είναι πραγματικά απαράδεκτο, δεν μπορώ να το ανεχτώ. Και δεν νομίζω ότι μπορούμε να αφήσουμε το Συμβούλιο να ξεφύγει με κάτι τέτοιο. Γιατί αλλιώ ε, παρεμποδίζεται η εκπροσώπηση των ε, πολιτών. Εμεί εκπροσωπούμε του πολίτες και οι πολίτες έχουν δικαίωμα να εκπροσωπούνται σωστά. Αν τώρα εμείς θέλουμε να εκπροσωπήσουμε σωστά τους πολίτες που μας εξέλεξαν, προφανώς πρέπει να έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίε. Δεν υπάρχει θέμα τέτοιο. Δεν μπορούμε να αποφασίσουμε για κάτι του οποίου το περιεχόμενο δεν γνωρίζουμε αν ένα αντικείμενο, αν ένα έγγραφο ε, δεν ε, μας δίδεται, σημαίνει ότι κάτι κρύβεται, ότι κάτι δεν έχει πάει καλά στο έγγραφο αυτό, ότι δεν πρέπει να βγει στη δημοσιότητα αυτό το κείμενο. Ε, αρχίζουν να δημιουργούνται εντυπωσει έτσι, δηλαδή κάτι δεν γίνεται, δεν συμβαίνει σωστά, δεν, κάτι δεν πάει καλά και γι' αυτό θέλει να κρατηθεί, θέλουν κάποιοι να κρατηθεί μυστικό. Ε, αυτό δεν νομίζω ότι μπορούμε να το πούμε. Ε, στην ε, Γερμανία η κοινή γνώμη γενικώ ε, ανησυχεί για την ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στη ζώνη Σέγγεν. Αλλά υπάρχουν αυτές οι ανησυχίες. Πώς θα τους καθησυχάσουμε εάν εμείς δεν έχουμε αυτές τις συγκεκριμένες πληροφορίες. Γιατί εγώ τώρα θα πάω στην πατρίδα μου και θα πω «Α, το Συμβούλιο δεν μας δίνει τις, τις πληροφορίες, ούτε μπορώ να τις δω» και η συγκήτρια μπορεί αλλά ε, μέσα στην ίδια ομάδα ακόμη μπορεί να, την πολιτική ομάδα μπορεί να υπάρχουν διαφορετικέ απόψει. Εγώ με, την, ε, με τον εισηγητή, εντάξει, τα πάω καλά στη συγκεκριμένη στιγμή, αλλά μπορεί να είναι κάποιο άλλο που να μην συμφωνούμε και να είναι διαφορετικέ οι απόψει. Και τι θα γίνει στην ψηφοφορία μετά. Δεν γίνεται να δώσουμε γνωμοδότηση χωρίς ο κάθε ένας από εμά να έχει πρόσβαση σε αυτά τα έγγραφα. Δεν γίνεται ή θα δώσουμε μια γνωμοδότηση που θα λέει ότι την απορρίπτουμε, γιατί δεν είχαμε πρόσβαση στα δεδομένα. Ίσως να μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό. Ε, όσο άκουγα το, το σκεφτόμουν. Ίσως θα μπορούσαμε ακριβώς γι' αυτό το λόγο να δώσουμε αρνητική γνωμοδότηση. Γιατί δεν μας δόθηκε πρόσβαση στα δέγγραφα. Και δεν μας αρνήθηκε η πρόσβαση από την Προεδρία, μας, την αρνείται το Συμβούλιο. Ίσως η Προεδρία δηλαδή να μην έχει και καθόλου λόγο όλο αυτό, δεν το ξέρω αυτό και δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά το Συμβούλιο γενικώ δεν θέλει να ως εκπρόσωποι εμεί των λαών να έχουμε άποψη για το τι περιλαμβάνουν αυτά τα έγγραφα. Ίσως λοιπόν να πρέπει να δώσουμε αρνητική γνωμοδότηση. Εάν δεν λάβουμε πρόσβαση σε αυτά τα έγγραφα. Χαίρομαι που ο πρόεδρο τη επιτροπή μα ε, ε, κινείται προ την ίδια κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Thank you, Mrs. Ernst. Ευχαριστώ κύριε Ernst. Σας ευχαριστώ. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστώ τον εισηγητή. Εγώ ως κοιόδης εισηγητριά συμμερίζομαι την άποψή σα και χαίρομαι που και ο πρόεδρο τη Επιτροπή μα ε, μίλησε ξεκάθαρα εγώ είμαι πάντα προσωπικά υπέρ του ανοιχτού λόγου, ίσως γι' αυτό δεν είμαι πολύ διπλωμάτη, αλλά τι να γίνει. Αλλά πραγματικά θα πρέπει να πούμε τα πράγματα έξω από τα δόντια, γιατί αλλιώ θα αφήσουμε να μα κοροϊδεύουν Εμά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και θα ήθελα να ρωτήσω, ποια είναι η βάση στον κανονισμό που βασίζεται ότι λέει ότι μπορεί να πάει ο συγητή και ε, οι συντονιστέ ξέρω εγώ, κάποιοι δεν ξέρω τι. Ποια είναι η βάση για κάτι τέτοιο. Θα ήταν ενδιαφέρον να το ρωτήσουμε. Μετά βέβαια να ρωτιέμαι τι μας αποκρύβουν, γιατί δεν μας δίνουν τα έγγραφα. Να ρωτήσουμε γιατί, γιατί και πώς το Συμβούλιο δημιουργεί μια τέτοια έλλειψη εμπιστοσύνη έναντι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και θέλω να σας πω και κάτι άλλο στα γερμανικά μέσα ενημέρωση μέχρι και το επίπεδο της, ε, των νομοσπονδιακών κρατηδίων γίνονται διάφορες εικασίες τι θα γίνει τώρα με τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία και την ένταξη στο Σέγγεν. Εγώ διάβασα στην εφημερίδα το Σαββατοκύριακο ότι η Γερμανία και η Γαλλία είναι κατάλογο διαφθοράς και επιδέλυψης της ασφάλειας αλλά και η Φιλανδία λέει είναι επίσης. Πολωνία και Τσεχία το σκέφτονται. Και στις 24 Φεβρουαρίου θέλει το Συμβούλιο να συμφωνήσει πάνω σε αυτά και θα δούμε μετά θα γίνει. Ε, υπάρχουν αυτές οι ανησυχίες και οι φόβοι των πολιτών που πρέπει να τράβει κανένα υπόψη, ιδίω όταν με ζει στα σύνορα και εκτό αυτού. Και δεν μπορούμε να απαντήσουμε. Και οι κασίες και οι κρατοσκοπίες αυτές γίνονται εις βάρος αυτών των δύο χωρών. Αυτό θέλω να τονίσω. Όλα αυτά είναι εις βάρος της εικόνες και της φήμης των δύο αυτών χωρών και δεν επιτρέπεται να δεχθούμε κάτι τέτοιο, νομίζω. Χαίρομαι για τις προτάσεις της κυρίας Φίμπερ και για αυτό που είπε και ο πρόεδρος της ομάδας της Επιτροπής μας. Θα πρέπει νομίζω να στείλουμε μια τέτοια επιστολή όπως εκείνη που ανέφερε η κυρία Βέμπερ να στραφούμε λέει προς το μέσω του κυρίου Μπούζεκ είναι νόμιμη αυτή η άγουσα και τελειώνω να σας πω ότι δεν θέλω επουδενή δεν θέλω να απαντήσουμε με μια αρνητική ψήφο. Γιατί αυτό δεν θα το καταλάβει στη Ρωμανία και Βουλγαρία κανεί. Να μην το κάνουμε. Αλλά να ζητήσουμε ξεκάθαρα να πάρουμε τα έγγραφα στα χέρια μα και να απαντήσουμε σωστά. Κύριε Λέντι Λάτφορντ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπαν οι συνάδελφοι. για τη διαδικασία και την έλλειψη των δικαιωμάτων ε, πρόσβασης των εκλεγμένων ε, ευρωβουλευτών. Όπως είπε η κυρία Βέιμπερ, συνανίστρια μας. Είναι απαράδεκτη η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Το μόνο που θέλω να πω και μην με παρεξηγήσετε Λέω ότι αυτή η έκθεση για την Ρουμπανία και τη Βουλγαρία θα πρέπει να εξεταστεί μέσα στα πλαίσια τη ε, νομική κατάσταση που ισχύει αυτή τη στιγμή. Ότι μπορεί δηλαδή να καλύψει μόνο τα θέματα που καταγράφονται στα πλαίσια διαδικασία ε, αξιολόγηση Schengen. Ταυτόχρονα όμω υπάρχει ο μηχανισμός ε, συνεργασίας και αξιολόγηση. Και δεν υπάρχει μια ε, εσωτερική νομική σχέση μεταξύ των δύο και γι' αυτό το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να μείνουν μέσα στα νομικά πλαίσια αυτής της διαδικασία. Αλλά μου φαίνεται με ένα περίεργο που δεν υπάρχει καμία αλληλένδεση μεταξύ των δύο. Και όχι μόνο τώρα σχετικά με την Ρουμανία και τη Βουλγαρία. Είναι σαν να φοράμε παροπίδες και εγώ μιλάω σαν υπήκος ε, μια χώρα που δεν είναι μέρος της διαδικασία Σέγγεν είτε το θέλω είτε δεν το θέλω αλλά μου φαίνεται περίεργο ότι μπορεί κανένα να μιλάει για την εφαρμογή των σωστών ελέγχων στα σύνορα αστυνόμησης ε, πρόσβαση στην ε, τράπεζα δεδομένων και να μιλάμε για εξασφάλιση της ε, δικαστικής ανεξαρτησίας, της καταπολέμησης της ε, διαφθοράς, ε, θέματα πρόσβασης των οργανωμένων εγκληματιών και αυτά να δεν σχετίζονται τα μεν με τα δε. Είναι γεγονό ότι έτσι έχει κατάσταση αυτή τη στιγμή. Και νομίζω ότι αυτό καταδεικνύει την περίεργη κατάσταση στην οποία έχει βρεθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ότι υπάρχει δηλαδή αυτό ο κατακαιρματισμό. Ενώ κατά βάση υπάρχουν αλληλενδέσεις μεταξύ των μεν και των δε. Δεν ξέρω αν σε αυτό αναφέρθηκε ο κύριο Κοέλια όταν στην έκθεσή του για την πρόσβαση στο σύστημα ενημέρωση του Σέγκερ αναφέρεται στην ανάγκη για ένα νέο σύστημα αξιολόγηση που θα πρέπει να είναι απλό, αποτελεσματικό και διαφανές και θα επιτρέπει να υπάρχει ο ελεύθερη κυκλοφορία στον χώρο Σέγγεν. Νομίζω θα πρέπει να ξανασκεφτούμε τι σημαίνει εποπτεία, αξιολόγηση, επιθεώρηση, επιβεβαίωση και ποιου τύπου χρειάζεται σε όλο τον χώρο Σέγγεν. Δηλαδή έχουμε τη συνδίκη της Λισαβόνας αλλά δεν έχουμε παρά ένα πεπαλαιωμένο σκεπτικό ότι δεν πρόκειται να κρίνουμε με τους δε. Δηλαδή, όπως το λέω εγώ, η νοοτροπία του διπλωματικού ομίλου. Αλλά η Βουλγαρία και η Ρουμανία πρέπει πραγματικά να κριθούν βάσει των πραγματικών νομικών προϋποθέσεων που ισχύει. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, εγώ σας ευχαριστώ. Ο Μαρινέσκου. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστώ τον κύριο Κοέλιο για την παρουσίαση που μας έκανε. και να σας ευχαριστήσω που βρήκατε μία λύση για κάθε ένα από τα σενάρια που προτείνονται, για κάθε μία από τις καταστάσεις που παρουσιάζονται. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω και όλους τους συναδέλφους. Συμφωνώ. Η ένταξη στον χώρο Σέγγεν θα πρέπει να δοθεί μόνο βάσει των εκθέσεων της ομάδας αξιολόγησης. Και επίσης η γνωμοδότηση του βινοβουλίου θα είναι πολύ σημαντική. Στην απόφαση 22 Ιανουαρίου θα υπάρχει συμπεράσματα της ομάδας του κ. Σαβά. Αυτά όλα θα πρέπει να ακολουθήσουν κάποιες ανακτικές που προτείνονται. Και μπορώ να συμφωνήσω ότι στις 3 θα υποβληθεί μια έκθεση και μετά σε μια έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής μας θα μπορούν να υποβληθούν τροπολογίες για να μπορέσουμε μετά να παρουσιάσουμε την έκθεση στην Ολομέλεια. Και έτσι θα έχουμε τη δυνατότητα να πάρουμε μια απόφαση που θα φασίζεται, επαναλαμβάνω, στα συμπεράσματα της ομάδας του κ. Σεβάν. Όσον αφορά την πρόσβαση στα έγγραφα, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Θα πρέπει να έχουμε πρόσβαση στα έγγραφα για να μπορέσουμε να αποφασίσουμε έγνωστα πραγμάτων. Η Ρουμανία και η Βουλγαρία ούτως ή άλλως ζήτησαν στο Συμβούλιο τα έγγραφα αυτά να μην θεωρούνται πια απόρριτα για να μπορέσει ακριβώς να επιληθεί αυτό το διοικητικό πρόβλημα. Τα μέτρα που πρότειναν οι συνάδελφοι περαϊφθούν τον γρηγορότερο δυνατόν, ούτω ώστε εμεί γρήγορα να έχουμε τι απαραίτητε πληροφορίε στα χέρια μα για να μπορέσουμε γρήγορα να πάρουμε μια απόφαση. Δεν θα ήθελα να αρνηθείτε για διοικητικού λόγους την ένταξη των δύο αυτοχωρών στον χώρο Σέγγεν. Δεν θα το καταλάβουν οι πολίτε των εν λόγω χωρών. Γιατί δηλαδή δεν θα μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω ε, μιας διαφοράς που υπάρχει μεταξύ δύο κοινοτικών θεσμικών οργάνων. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να λύσουμε αυτά τα ε, προβλήματα, ιδίως αν δεν μπορέσουμε να βρούμε ένα συμβασμό. Επαναλαμβάνω, η Ρωμανία και η Βουλγαρία ζήτησαν την άρση του απορρίτου των εγγράφων αυτό και να μπορούμε να το γνώσουμε λόγω των δυνατών. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κυρία Στανόκα. Thank you, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, παίρνω τελευταία το λόγο, παρόλο που... Όχι, δεν θα είστε τελευταία. Έχουμε και άλλους. Οπότε, επειδή έχουμε και άλλους, να σας θυμίσω να είστε σύντομοι και να μείνετε στην ουσία του πράγματος για να προχωρήσουμε γιατί έχουμε κι άλλο ένα σημείο να συζητήσουμε. Ναι, αλλά οι σκιώδες συνήθω μιλάνε πρώτοι. Μπας Εγώ απλώς θέλω να πω ότι μπορώ να εξάγω συμπέρασμα ότι είμαστε ομόφωνοι στο θέμα αυτό, που είναι σπάνιο. Νομίζω ότι είναι το αντίθετο από αυτό που ήθελε τελικά το Συμβούλιο από το Κοινοβούλιο. Και τώρα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε αυτό που προτείνει ο εισηγητής. Και χαίρομαι που είναι σαφής η έκθεσή του και χαίρομαι και για τις επιστολές που αποστήλατε εσείς Πρόεδρε δείχνοντας τη σαφή μας θέση για την πρόταση του Συμβουλίου. Εγώ δεν θα είχα ε, ε, πρόσβαση σε αυτά τα έγγραφα ούτως ή άλλως, γιατί είμαι και σκιώδης συζητήτρια από τους πράσινους και Νομίζω ότι σε ό,τι αφορά την ζώνη Σέγγεν και την ένταξη της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας, ε, ότι θα πρέπει όντως να ενταχθούν οι δύο αυτές χώρες. Χωρίς να υπάρχουν προκαταλήψεις. Δεν θέλω να μακρηγορήσω γιατί τα περισσότερα υπόθηκαν. Να πω απλώς ποια είναι η θέση των πρασίνων. Εμείς υποστηρίζουμε Πλήρω την ε, γνωμοδότηση του εισηγητού. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Πάντα προσπαθούμε να δώσουμε προτεραιότητα στους σκιώδεις εισηγητές, να μιλούν πρώτοι. Αλλά ε, δεν τα καταφέρνουμε και πάντα. Υπήρχαν ε, δυο σκιώδεις πέραν του κυρίου Κοέλιο αλλά να ξέρετε ότι πάντα προσπαθώ να σας βάζω να μιλάτε πρώτοι. Ο κύριος Κλέης έχει το λόγο. Αν θέλετε να είστε σύντομος γιατί έχουμε μεγάλο κατάλογο. Δεν θα μιλούσα όσο οι προηγούμενοι. Ο κύριος Κοέλιος στην παρουσίαση το έχει απόλυτο δίκιο. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να περάσει αυτό που θέλει το Συμβούλιο. Είμαστε μέλη του Κοινοβουλίου και πρέπει να έχουμε λόγο. Ε, επίσης αυτή η πρόταση που έκανε εσύ Πρόεδρε για το Κοινοβούλιο ότι θα πρέπει να ζητήσουμε από το Συμβούλιο να, έχει, να έχουν πλήρη πρόσβαση όλα τα μέλη της Επιτροπής του Κοινοβουλίου ε, στα έγγραφα αυτά. Εάν δεν μπορούμε να μάθουμε όλη την αλήθεια, προφανώς θα υπάρξουν προβλήματα. Υπάρχουν διάφορες φήμες που κυκλοφορούν, που λένε ότι μια χώρα συμφωνεί, μια χώρα, δεν είναι, μια χώρα είναι εντάξει, μια χώρα δεν είναι. Ε, αλλά πρέπει αυτό να μπορούμε να το αποδείξουμε επί τη βάση επισήμων εγγράφων. Υπάρχουν και, υπάρχει και ένα κοινό μνημόνιο ε, της Europol, της Eurojust ε, ε, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, που αναφέρεται εκεί, αναφέρονται τα προβλήματα που υπάρχουν στην, στην Βουλγαρία και τη Ρουμανία, ειδικά Μάλλον όχι ειδικά για τη Σέγγεν, αλλά υπήρχαν κάποιες στοιχείες που αφορούσαν και την ζώνη Σέγγεν. Αλλά αν δεν έχουμε εμεί πρόσβαση για να δούμε τι λένε αυτά τα έγγραφα, νομίζω ότι θα πρέπει να καταψηφίσουμε, να δώσουμε αρνητική γνωμοδότηση για όλη την πρόσβαση της ε, Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. Um, Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή και όλους τους συναδέλφους για την υποστήριξή σας για την ε, προσχώρηση της Ρουμανίας και της ε, Βουλγαρίας στο χώρο Σέγγεν. Θα ήθελα να αποβάλω τέσσερις ε, σύντομες ερωτήσεις σε σχέση με το CVM, γιατί ε, από όσο γνωρίζω και η κυρία Λάτφορτ ασχολήθηκε με αυτό το θέμα. Μιλάμε για ένα σύγχρονο μέσον που θα βοηθήσει αυτές τις χώρες έτσι ώστε να προωθηθεί και η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς. Αλλά δεν θα πρέπει να αποτελέσει πρόκριμα. Εγώ ήμουν υπουργό δικαιοσύνης όταν επινοήθηκε αυτός ο μηχανισμός τον χρησιμοποιήσαμε και θα τον χρησιμοποιούμε και στο μέλλον. Δεύτερον, θα πρέπει κατηγορηματικά να έχουμε πρόσβαση στις τεχνικές αυτές αποτιμήσεις έτσι ώστε να μπορέσουμε να αποφασίσουμε. Δεν μπορούμε να αποφασίσουμε χωρίς τις τεχνικές αυτές, ε, τα τεχνικά αυτά τα στοιχεία για μια χώρα η οποία έχει μια θετική αποτίμηση δεν υπάρχει λόγος αναβολής. Γιατί έγινε αυτός ο συσχετισμός και γιατί υπάρχουν τεχνικές αξιολογήσεις αν δεν λαμβάνονται υπόψη στην τελική απόφαση. Θα πρέπει να μπορούμε να εκφράσουμε και την κοινή γνώμη στις δύο αυτές χώρες και στα άλλα κράτη-μέλη να εξηγήσουμε γιατί λαμβάνουμε αυτή την απόφαση. Θα πρέπει να προβάλλουμε συγκεκριμένα επιχειρήματα και τέλος θα ήθελα να κρατήσουμε το τρέχον χρονοδιάγραμμα έτσι ώστε το Μάρτιο να μπορέσουμε να προσχωρήσουμε. Γνωρίζουμε ότι θα πρέπει να έχουμε πρόσβαση στα έγγραφα και είμαστε αλληλέγγυοι ως προς το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Χολμάιερ. Ναι, ε, πρόεδρε, εγώ ε, είμαι από μια περιφέρεια η οποία είναι στα σύνορα με την Τσεχία και έχουν ε, γίνει πολλές συζητήσει για το πόσο καταστροφικό ήταν το άνοιγμα των συνόρων και το πώς, ε, ε πώς έγινε η ένταξη της Τσεχίας στην Σέγγεν. Ε, βεβαίως τώρα έχουμε λιγότερα ε, εγκλήματα από παλαιότερα και ε, έχει, έχουν συνηθίσει οι άνθρωποι. Οπότε πρέπει να δείξουμε και την θετική πτυχή του να μπαίνει κάποιο στην ζώνη Σέγγεν. Ε, Συμμερίζομαι βεβαίω ε, πλήρω την άποψη του εισηγητού ότι τα έγγραφα όντως θα πρέπει να μας δοθούν, να πρέπει να δημοσιευθούν. Μιλούμε για ασφάλεια. Ε, νομίζω ότι απλώς τα κράτη-μέλη δεν έχουν συνηθίσει ακόμη να χρησιμοποιούν ή δεν έχουν συνηθίσει ότι ισχύει η, η Λισαβόνα. Εγώ υποστηρίζω απόλυτα την επιστολή και επίσης να πω σαφώς ότι δεν, μπορούμε να μας δεν μπορούν να μας βάζουν τους εισηγητές και τους σκιώδεις σε τέτοια α, δύσκολη θέση ε, να μας δίνουν μεν κάποιε πληροφορίες και μετά να μην μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε, να μην μπορούμε να τις συζητήσουμε. Ε, θέλουμε να εκπονήσουμε μία γνωμοδότηση. Ε, δεν γίνεται να μην ε, συζητήσουμε, ούτε να μην συζητήσουμε γίνεται, ούτε να μην έχουμε πλήρη δεδομένα γίνεται. Για τον εισηγητή ε, ο εισηγητή μπαίνει σε πολύ δύσκολη θέση, σε αδύνατη κατάσταση. Δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι. Νομίζω λοιπόν ότι για κάποιους τομείς ε, δεν θα πρέπει να προχωρήσουν κάποιες ε, καταστάσεις που έχουν ξεκινήσει και νομίζω ότι αυτό είναι ένας από αυτούς τους τομείς. Ελπίζω το Συμβούλιο να έρθει στα λογικά του η συμφωνία Σέγγεν πρέπει να ισχύει ή να είναι ίδια και με αυτούς που είναι μέλη της Σέγγεν και με αυτούς που θέλουν να μπουν στη Σέγγεν. Αν υπάρχουν τώρα επιπλέον ε, κριτήρια ε, τα οποία ανησυχούν κάποιους, θα πρέπει το Συμβούλιο να τα πει. Σαφώς και ξεκάθαρα. Θα πρέπει αυτά να είναι γνωστά. Θα πρέπει να πληρούνται από όλους. Και ε, χαιρετίζω αυτό που είπε στην Ολομέλεια ο Κάρλος και νομίζω ότι θα πρέπει να το ξανασκεφτούμε και εδώ, μήπως θα μπορούσαμε στα πλαίσια της συμφωνίας της Σέγγεν να δούμε, να αξιολογήσουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα και την, ε, το τι έχει γίνει με τα κράτη-μέλη που είναι ήδη α, ε, ε, μέλη της Σέγγεν. Δηλαδή εκ των υστέρων να γίνεται μια αξιολόγηση το αν πληρούνται τα κριτήρια. Η Βουλγαρία και η Ρουμανία τώρα νομίζω ότι πρέπει να έχουν και μια απόλυτη σαφήνεια για το τι πρέπει να γίνει με την περίπτωσή τους να μην δημιουργούμε μόνο ε, ανησυχίες, ούτε σε αυτές τις δύο χώρες που θέλουν να μπουν, ούτε στις χώρες που είναι ήδη μέλη, γιατί δημιουργούνται φόβοι και ε, καταστάσεις που ούτως ή άλλως στην πραγματικότητα δεν υφίστανται. Ευχαριστώ. Η κυρία Γιώτοβα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συγχαρητήρια στον εισηγητή Κοέλιο για το πώς χειριστήκε το θέμα με, την, με το Συμβούλιο και που μελέτησε διάφορες εναλλακτικέ για το πώς μπορούμε να προχωρήσουμε. Σε αυτά που υπόθηκαν να προσθέσω και εγώ κάτι. Είναι δύσκολο. Είναι, η δική μου χώρα, η Βουλγαρία, είναι σε μια ενδιάμεση κατάσταση αυτή τη στιγμή. Και μιλώ και ως μέλος της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ, αλλά και ως Βουλγάρα υπήκος. Είχαμε ζητήσει επισήμως από την, ε, την ε, επισήμω τα έγγραφα αυτά για την αξιολόγηση Σέγγεν από την ομάδα αξιολόγηση Σέγγεν Στι 21 Δεκεμβρίου το η Κομισιόν ήδη είχε λάβει την επιστολή από τη Γαλλία και τη Γερμανία που έλεγε ότι η ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας θα πρέπει να ε, αναβληθεί και θα πρέπει να πληρούνται τρία νέα τεχνικά κριτήρια. Και αυτό μας έδωσε την εντύπωση ότι υπήρχε, ήταν προαποφασισμένο αυτό. Ε, λυπούμε, συνάδελφοι, αλλά όλη αυτή η συζήτηση που γίνεται τώρα και με όλα όσα γίνονται στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα φαίνεται ότι είναι τελείως άχρηστε. Γίνεται πολλή συζήτηση και στα ΜΜΕ ε, και, στις, ε, και στη χώρα μου αλλά και στη Ρουμανία για τα ε, πρότυπα αυτά γιατί δεν είναι πολύ μακρινά το παρελθόν που έγιναν και άλλε χώρε μέλη στη Σέγγιν και τότε δεν υπήρχαν αυτά τα επιπλέον κριτήρια. Να σα θυμίσω ότι το Φλεβάρι αναμένεται τεχνική έκθεση για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία που θα λέει ποια είναι η πρόοδος για τους ε, μηχανισμούς ε, πιστοποίησης και, και ε, συνεργασίας. Νομίζω λοιπόν ότι ότι θα πρέπει να υποστηρίξουμε πλήρως, εγώ υποστηρίζω πλήρως πάντως, την σύνταξη της επιστολής μετά από με πρωτοβουλία του κυρίου Μπούζεκ και το θέμα αυτό πρέπει να λυθεί στο ανώτατο δυνατό επίπεδο. Γιατί αυτή η κατάσταση προκαλεί σχόλια, φήμες και όποιο ενδιαφέρεται στην, ε, για την ένταξη της ε, Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στη Σέγγεν δεν ενδιαφέρεται καθόλου για την, για την ε, τήρηση αυτών των κριτηρίων που επιχάρτω χάρτου υπάρχουν αλλά ουσιαστικά είναι θέμα πολιτική βούληση. Οπότε τι ακριβώς λέμε εδώ, ότι ε, γίνεται κάποια, κάποια, ως, ε, κατα, κάποια κατανομή ισχύω και αρμοδιοτήτων. Μπορώ να συζητήσουμε πολλά πράγματα για το θέμα αυτό, αλλά νομίζω ότι πρέπει να επανέλθουμε στα βασικά, ότι οι δύο αυτές χώρες είναι έτοιμες σε σχέση με τα τεχνικά κριτήρια για να γίνουν μέλη της Schengen. Εγώ υποστηρίζω αυτό που λέει ο κύριο Κοέλιο, να μην δώσουμε γνωμοδότηση πριν λάβουμε πλήρες πληροφορίες για τα έγγραφα αυτά, γιατί αλλιώς θα, κάνουμε, θα λάβουμε μια απόφαση η οποία δεν θα είναι βασισμένη σε τίποτα ουσιαστικά. Ε, Φαίνεται ότι υπάρχει ένα πρόβλημα Υπάρχει μια διαδικασία στο Συμβούλιο, στο Συμβούλιο μια διαδικασία στο Κοινοβούλιο, αλλά φαίνεται ότι δεν τηρούνται. Αυτό αφορά το θέμα των τεχνικών στοιχείων που χρειαζόμαστε για την εκθεσή μας και τη δυνατότητα πρόσβαση. Άκουσα προσεκτικά αυτά που είχαν να πούνε οι συνάδελφοι από την χώρα προέλευσής τους. Φαίνεται ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια τάση για την τοποθέτηση διαφόρων κρατών μελών. Στην αφορά τη θέση του κυρίου Κοέλιο, που έχει δυνατότητα πρόσβαση σε περισσότερε πληροφορίε από εμά, θεωρώ ότι θα πρέπει πραγματικά να πιστέψουμε τον εισηγητή μας και αντίθεση από αυτά που λένε οι συνάδελφοι δεν νομίζω ότι θα πρέπει να καταψηφίσουμε αν δεν έχουμε επαρκή ψηφοφορίες γιατί εδώ πρόκειται για μια δημοκρατική διαδικασία που θα πρέπει να εφαρμόσει κατά τον ίδιο τρόπο όλων σε όλες τις χώρες μέλη του Σέγγεν και δεν μπορούμε να εισαγάγουμε εδώ νέες κανόνες κατά διάρκεια διαδικασίες. Αυτό δεν νομίζω ότι σχετίζεται με τους πολύ συγκεκριμένους όρους που, θα, που ισχύουν για τη δυνατότητα ένταξη των χωρών Σέγγεν. Τώρα, πώς θα εξηγήσουμε την κατάσταση στους πολίτες είτε είναι πολίτες των παλιών ή των νέων χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να τους εξηγήσουμε τι είναι ο χώρος Σέγγεν, ποιοι είναι οι όροι που πρέπει να πληρώνουν και να τους πούνε τα πράγματα ξεκάθαρα και να χρησιμοποιήσουμε την ίδια δημοκρατική διαδικασία για να το κάνουμε. Και γι' αυτό θεωρώ ότι καταρχήν πρέπει να δώσουμε απόλυτη εξοπιστία στον εισηγητή κύριο Κοέλιο, να τον πιστέψουμε για το πώς θα πρέπει να ψηφίσουμε την έκθεση αυτή. Δηλαδή δεν ξέρω γιατί θα πρέπει να καταψηφίσουμε και θεωρώ ότι θα πρέπει να ασκήσουμε πίεση στο Συμβούλιο για να μπορέσουμε το γλυκότερο να τον έχουμε πρόσβαση σε αυτά τα έγγραφα. Ευχαριστώ κύριο Ποστινάρο. Thank you Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα μου επιτρέψετε να μιλήσω ρουμανικά. Εγώ είμαι μέρο ε, τη ε, αντιπολίτευση ε, στην Ρουμανία και επικρίνω συνεχώ το καθεστώς στην Ρουμανία. Αλλά εγώ τώρα δεν μιλάω ως Ρουμάνος, αλλά μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και βλέπω διάφορα πράγματα. Καταρχήν, τα κριτήρια εφαρμόζονται σε άλλα κράτη-μέλη της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν εντάχθηκαν στη, στο χώρο Σέγγεν. Αυτά τα κριτήρια άλλαξαν τότε χωρίς να το πει κανένας Ή προτίθεται ίσως να αλλάξουν οι κανόνες αυτοί. κατά βάση ένας κανόνας της νομοθεσίας είναι ότι οι νόμοι δεν μπορούν να ισχύουν αναδρομικά. Αν αλλάξουν τα κριτήρια δεν μπορούν να εφαρμοστούν παρά για τις μελλοντικέ διαδικασίες, όχι αυτές που αυτή τη στιγμή βρίσκω εδώ. Για την Ρουμανία και την ε, Βουλγαρία ισχύουν λοιπόν ήδη οι κανόνες που ισχύουν και για τις άλλες χώρες όταν εντάχθηκαν στο χώρο Σέγγεν. Ορισμένε από τι δηλώσει που έγιναν στο Βουκουρέστι είναι απαράδεκτε. Ναι, αλλά εδώ δεν ζητάμε για δηλώσει. Δεν πρέπει να συγχαίουμε τι ε, δηλώσει αυτές με την ρήτρα συνεργασία και εποπτεία. Άλλο αυτό. Άλλο τα κριτήρια ένταξης στο χώρο Σέγγεν τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να πάρουν απόφαση για την ένταξη στον χώρο Σέγγεν παρά πα, βάσει αυτών των κριτηρίων που ισχύουν. Χαίρομαι λοιπόν με τη θέση του κυρίου Κοέλιο, του εισηγητή μας και σας ζητώ να προσαντουστούμε απόλυτα με τα έγγραφα αυτά και να σεβαστούμε τους κανόνες που έχουν υιοθετηθεί. Και η ψηφοφορία που θα γίνει θα πρέπει να βασίζεται πάνω τα συμπεράσματα τη τεχνική έκθεση και όχι πάνω σε πολιτικέ ε, δηλώσει που δεν έχουν καμία σχέση με το χώρο Σέγγεν. Ευχαριστώ κύριε Μελίτεβα. Ευχαριστώ και εγώ θα ήθελα με τη σειρά μου να υποστηρίξω τον συνάδελφο Κάρλος Κοέλιου και όλα όσα προελέχθησαν από τους συναδέλφους έτσι ώστε όλοι οι ευρωβουλευτές να έχουν τα στοιχεία αξιολόγησης για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία και αυτό είναι και προς ε, το συμφέρον του Συμβουλίου για να υπάρξει πλήρης διαφάνεια και να μην υπάρξει οποιαδήποτε εικασία επί του θέματος όπως ισχύει σήμερα. Διαφορετικά συγχαίουμε τα πάντα. Η Γαλλία και η Γερμανία ε, μιλάν συγκαλυμμένα για πολιτικούς λόγους. Αλλά δεν μιλούν για τα τεχνικά κριτήρια τα οποία θα πρέπει να πληρεί κανείς για να μπορέσει να μπει στο Σέγγεν. Θα ήθελα το Συμβούλιο να δώσει στο Κοινοβούλιο αυτά τα στοιχεία και η Γαλλία και η Γερμανία θα πρέπει να μας δώσουν πιο ε, συγκεκριμένα στοιχεία. Γιατί δεν θέλουν την προσχώρηση, δηλαδή αναμένουμε δύο μηνύματα από το Συμβούλιο. Καταρχήν να υπάρξει διάλογος και συνεργασία μεταξύ όλων των θεσμικών οργάνων και να δούμε την όλη διαδικασία έτσι ώστε να μην υπάρχει έλλειψη διαφάνειας και να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό, αυτά τα δεδομένα για τις μελλοντικές αποφάσεις. Αυτό αφορά την αξιοπιστία μας έτσι ώστε όλοι οι πολίτες και οι Ρουμάνοι και οι Βούλγαροι να πιστεύουν σε μας. Ευχαριστούμε πολύ. Είχαμε πολλές παρεμβάσεις. Δεν βλέπω να υπάρχουν άλλοι βουλευτές που θα ήθελαν να παρέμουν. Κύριε Έντσιου, θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο ή διαδικαστικό. Θα ήθελα. Τώρα το σκέφτηκα. Να σας πω το εξής επειδή πρόκειται για μια κατάσταση χωρίς προηγούμενο που δημιουργήθηκε με το Συμβούλιο να συμβουλευτούμε τη νομική μας υπηρεσία και αν μας το αρνηθούν να μπορέσετε να κάνετε προσφυγή στο ΔΕΚ κατά του Συμβουλίου γιατί θα πρέπει να τηρηθεί το γράμμα της Συνθήκης της Λισαβόνας. Ευχαριστώ. Αυτό θα έλεγα και εγώ υπενθυμίζοντας ότι έχει μεγάλη σημασία η πρόσβασή μας πριν ε, λάβουμε μία απόφαση, διότι αυτό είναι και καθήκον μας ως προς το θέμα αυτό. Όχι μόνο για να ε, πληρωθεί το γράμμα της συνθήκης της ε, Λισαβόνας, ως προς να αγαστεί συνεργασία δηλαδή μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου, αλλά και επειδή είναι θέμα αρχής και σεβασμού προς εμάς. Πέρα από την ε, ουσία του θέματος, νομίζω ότι υπάρχει μία μεγάλη συνένεση που υποστηρίζει την ε, επέκταση του κεκτημένου του Σέγγεν ως προς την ουσία του θέματος. Αλλά ως θέμα αρχής θα ήθελα να ερμηνεύσω αυτή, αυτό το στοιχείο, ότι δηλαδή θα αποστείλουμε μία επιστολή στο Συμβούλιο, διότι στη Βουδαπέστη, στο Συμβούλιο Υπουργών, κατά τις τελευταίες, όπως έγινε και κατά τις τελευταίες μέρες της ε, Βελικής Προεδρίας, έτσι κάνουμε και τώρα, υπό Ουγγρική Προεδρία, δηλαδή θα αποστείλουμε μια επιστολή στο Συμβούλιο ερμηνεύοντας το πνεύμα αυτών των δεδομένων μετά από την ε, σε έκταση συζήτηση που έγινε, έτσι ώστε να δούμε ποια θα ήταν τα ενδεχόμενα επιπρόσθετα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν. Αύριο το πρωί θα γίνει μια συνάντηση των συντενιστών. και θα δούμε κατά πόσο θα πρέπει να προσφύγουμε στη νομική υπηρεσία και να προωθήσουμε, να προβάλλουμε το δικαίωμά μας να ασκήσουμε προσφυγή ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου έτσι ώστε να τηρηθεί το γράμμα της συνθήκης της Λισαβόνας ως προς συνεργασία μεταξύ Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διότι νομοθετούμε από κοινού. Και θα ακολουθήσουμε το χρονοδιάγραμμα όπως ορίστηκε και θα ακούσουμε και τι θα έχει να μας πει ο κύριος Κοέλιου. Νομίζω ότι σας υποστήριξαν οι πάντες κύριε Κοέλιου. Θα ακούσουμε την Επιτροπή Ίσως η Προεδρία θέλει κάτι να πει. Η Προεδρία, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Κατά τη διάρκεια του πρωινού, το θέμα της πρόσβασης των εγγράφων ακούστηκε και δεν μπορώ παρά να επαναλάβω αυτή τη θέση πρόσβαση στα έγγραφα. Ε, έχουμε πληροφορηθεί σε σχέση με το αίτημά σα και τη σημασία του. Επίπεδο Συμβουλίου καταβάλουμε κάθε προσπάθεια έτσι ώστε να ανταποκριθούμε στο αίτημά σα, το οποίο είναι καθόλου νόμιμο υπό την ίδια έννοια δεν μπορούμε παρά να λάβουμε υπόψη και τον κανονισμό λειτουργίας του Συμβουλίου. Θα εξέπρουμε μία λύση έτσι ώστε να έχετε και το περιεχόμενο, σας γνωστοποιηθεί και το περιεχόμενο αυτή της έκθεσης. Η Επιτροπή θα ήθελε να μιλήσει. Όχι. Δεν έχουμε ε, συγκεκριμένο, λάβει συγκεκριμένο έργο ως προς την ε, προσχώρηση στο χώρο του Σέγγεν. Άρα δεν έχουμε κανένα σχόλιο, λέει η Κομισιόν ε, Κοέλιου. Ο κύριος Έντσιου έχει απόλυτο δίκιο. Θα πρέπει να γίνει μία συνάντηση για να λάβουμε υπόψη την στρατηγική μας. Αύριο στις 4 προτείνω να συναντηθούμε με τους σκιώδεις. Δεν θα γίνει μακρά συζήτηση, αλλά τουλάχιστον να μπορέσουμε να εργαστούμε. Θα σας στείλουμε, θα στείλω ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για όλους τους σκιώδεις. Κάποιος ε, ρώτησε γιατί έχουμε τέτοιο, τέτοια προβλήματα με τα έγγραφα της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. Και μας εξέπληξε η απάντηση γιατί μας ελέγχθη ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με τη Ρουμανία και τη Ρουμανία, αλλά δεν θέλει το ε, Συμβούλιο να δημιουργηθεί προηγούμενο. Δηλαδή, μια τέτοια διαδικασία θα προβάλλουμε και σε άλλες περιστάσεις παρόμοιες. Ε, δεν αφορά τις δύο αυτές χώρες, αλλά θέληση του Συμβουλίου είναι να μην δώσει τα έγγραφα αυτά σε όλες τις παρόμοιες υποθέσεις και αυτό είναι ακόμα πιο σοβαρό. Τρίτον, θα συνεχίσω στα αγγλικά. Ορισμένοι συνάδελφοι πρότειναν το εξής, επειδή είμαστε θυμωμένοι με το Συμβούλιο, να αποφανθούμε αρνητικά. Δεν ε, συμμερίζομαι αυτή την άποψη, διότι η Ρουμανία και η Βουλγαρία δεν μπορούν να είναι ε, θύματα μίας θεσμικής διένεξης μεταξύ των δύο οργάνων. Εάν ε, παραταθεί αυτή η διαδικασία, προτείνω να μην επιτρέψουμε στο Συμβούλιο να πει ότι δεν θα αποφανθεί τελικά, διότι περιμένει τη Συμβουλή του Κοινοβουλίου. Δηλαδή μπορούμε να προβούμε σε μία γνωμοδότηση λέγοντας ότι επειδή δεν μας δόθηκαν τα έγγραφα δεν θα μπορέσουμε να γνωμοδοτήσουμε. Από νομικής πλευράς γνωμοδοτούμε αλλά χωρίς περιεχόμενο. Τέλος. Η Βαρόνι Λάντφορτ έκανε ένα πολύ ενδιαφέρον σχόλιο σε σχέση με το σύστημα Σέγγεν. Θα θυμόσαστε μερικοί ότι είχα πει ότι τις πρώτες πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα έπρεπε να, τις, να μην τις ε, λάβουμε υπόψη και η Επιτροπή Μπαρόζο 2 προέβαλε ένα νέο σύστημα. Uh, ένα νέο σύστημα αξιολόγησης. Και πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουμε την συναπόφαση Δηλαδή θα εισακουστεί η άποψη του Κοινοβουλίου από το Συμβούλιο διότι συνομοθετούμε. Και νομίζω ότι η κυρία Λάτφορντ έχει δίκιο γιατί η συζήτηση για το νέο σύστημα αξιολόγησης είναι ο κατάλληλος ο χώρος για να αντιμετωπίσουμε ορισμένα τα ζητήματα που μας απασχολούν. Και κάτι μας είπε η Μόνικα Μάιερ Είπα και στην Ολομέλεια ότι το σύστημα που έχουμε τώρα δεν είναι το καλύτερο δυνατό. Αυτοί που ήδη συμμετέχουν ίσως είναι πολύ αυστηρές για αυτούς που θέλουν να προσχωρήσουν και είναι ιδιαίτερα νοθρές για αυτούς που ήδη βρίσκονται στο σύστημα Σέγγεν. Αυτό που έχει σημασία λοιπόν είναι να αντιμετωπίσουμε τις χώρες ισότιμα και δίκαια, δηλαδή ο, οι ίδιοι κανόνες να ισχύουν για όλους. Και θα γίνει η συζήτηση, η πρώτη ανταλλαγή απόψε την επόμενη εβδομάδα στις 31 Ιανουαρίου για το νέο σύστημα αξιολόγησης. Ευχαριστούμε κύριε Κουέλιο. Πολλά ουσιώδη σημεία αναφέρθηκαν και αύριο θα δούμε στους συντονιστές τι μέσα έχουμε στη διάθεσή μας για να επιβεβαιώσουμε αυτούς τους, αυτά τα ζητήματα αρχής τα οποία θίξαμε, δηλαδή να ληφθεί υπόψη η άποψη του Κοινοβουλίου, να ληφθεί πλήρως η άποψη του Κοινοβουλίου, όπως και σε άλλα συναφή ζητήματα που θα ανακύψουν στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ και πάμε στο επόμενο θέμα.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 If you please, those who stay in the room remain silent. help. Παρακαλώ λίγη ησυχία στη αίθουσα για να περάσουμε στο σημείο περιθμών 10. Τελευταίο σημείο για σήμερα. που το 6 και το 7 θα εξεταστεί αύριο. Το σήμα 10 αφορά κυκλοφορία στην αγορά και χρήση πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών. Και ο εισηγητής είναι εδώ, ο συνάδελφος Γιάνν Μούλτερ. Ο στόχος είναι να ακούσουμε την παρουσία της Κομισιόν αυτή τη στιγμή. Γιατί πρόκειται για μια πρόταση της Κομισιόν. Κυκλοφορία στην αγορά και χρήση προδρόμων εκλεκτικών υλών. Και ο στόχος είναι να μειωθεί η πρόσβαση του κοινού σε χημικές ουσίες υψηλού κινδύνου που μπορούν να βοηθήσουν στην παραγωγή εκλεκτικών υλών. Θα ακούσουμε λοιπόν πρώτα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας τοποθετήσει μέσα στην πρόταση και μετά θα ακούσουμε τον εισηγητή Γιάνν Μιούλτερ και τα άλλα μέλη που θέλουν να κάνουν δηλώσεις. Πρώτα λοιπόν ο εκπρότωσος της Κομισιόν. Κύριο Σίφερ. Uh, Ευχαριστώ πρόεδρε. Καλησπέρα κύριε και κύριοι. Μπορεί να είμαι πάρα πολύ σύντομο. Γιατί η πρόταση που έχω να σας παρουσιάσω σε γενικές γραμμές είναι πάρα πολύ τεχνική, αλλά εξ αυτού και πολύ σαφής. Ευνόητη και απλώς συνεχίζει ένα πρόγραμμα δράσης της Κομισιόν του 2008 που αυξάνει την ασφάλεια των εκλογικών υλών. Λοιπόν, θέλουμε να υπάρχει περιορισμένη πρόσβαση στις χημικές αυτές ουσίες και ο στόχος είναι να μειωθεί κατερχήν η απειλή τους πολίτες από τα αποτελέσματα αυτών των ε, κρυκτικών υλών και δεύτερον να δημιουργεί ένα ίσο πεδίο δράσης στους παραγωγούς ούτω ώστε να είναι σίγουρο ότι στην εσωτερική αγορά δεν θα υπάρχουν στρεβλώσει λόγω διαφορετικών κανονισμών ασφαλεία που εφαρμόζονται στα διάφορα κρατημέλη. Η πρωτοβουλία αυτή που σας είπα είναι μία από τις 50 δράσεις του προγράμματος δράσης της Κομισιόν του 2008 το υπόβαθρο λέω είναι ότι οι περισσότερες um, οι περισσότερες τρομοκρατικές οργανώσεις χρησιμοποιούν αυτού του είδους τις ουσίες. Αυτές οι χημικές ουσίες με τις οποίες μπορούν να κατασκευάσουν κριτικές ε, ύλες και οι οποίες είναι ευρέως διαθέσιμα στο ευρύ κοινό. Και γι' αυτό η προτινόμενη άουσα από την Κομισιόν είναι να απαγορευτούν οι σημαντικότερες αυτές τις πρόδρομες ουσίες για την χρήση από το ευρύ κοινό και σε ένα παράρτημα της ε, οδηγίας να αναφέρονται αυτές οι ουσίες και να αναφέρεται επίσης ένα κατόφλιο συγκέντρωσης ποσοτικό κάτω από το οποίο δεν είναι επικίνδυνες και μπορούν να πολιθούν στο ευρύ κοινό. Πάνω από το κατόφλιο μας αυτό θεωρούνται ιδιαίτερα επικίνδυνες και γι' αυτό δεν θα πολλούνται στο ευρύ κοινό. Ο κανονισμός που ισχύει αυτή τη στιγμή um, δεν θα ισχύει στις ε, συναλλαγές ε, επιχειρήσεων και δεν θα αφορά προσμίξεις που χρησιμοποιούνται από τις στρατιωτικές δυνάμεις ή δυνάμεις επιβολής του νόμου. Ο στόχος είναι ακριβώς το ευρύ κοινό και η ανάγκη δημιουργίας ε, κάποιων μέτρων για τους ε, εμπόρους. Ο κατάλογος αυτός θα πρέπει να ενταχθεί ε, όπως σας είπα μέσα στα πλαίσια των δράσεων για το, που απορρέουν από το πρόγραμμα του 2008 και αποτελείται από εμπειρογνώμονες ασφαλεία από τα κράτη-μέλη, η Εν Επιτροπή, από εκπροσώπους Βιομηχανία. Το συζητήσαμε διαμακρών, εμπιστευτικά, έχουν τεθεί δηλαδή όλα τα χαρτιά επί τάπητος. Έχουμε τεχνικές και επιστημονικές γνωμοδοτήσεις όσον αφορά το κατόφλι στο οποίο θα πρέπει να έχουμε στους ποσοτικούς περιορισμούς. Μερικές από αυτές τις ουσίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα από τρομοκράτες. Αυτές δεν έχουν όμως αναφερθεί στον κατάλογο γιατί είναι τόσο ευρέως δεδομένοι που μία απογόρευση δεν θα μπορούσε αποδεισματικά να ελεχθεί. Παραδείγματο χάρη σκόνη αλουμινίου που μπορεί τόσο εύκολα να παραχθεί. Δεν αναφέρεται στον κατάλογο αυτό. Οι όλες ουσίες όμως που αναφέρουμε καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι είναι επικίνδυνες πέρα από τα κατόφλα αυτά και ότι η απογόρευσή τους θα μπορούσε να κάνει σημαντική και σαφή διαφορά στο μέλλον. Αυτό μέσα βέβαια για να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί πρέπει να προσαρμοστεί μέσω μιας διαδικασίας ε, διευκολυνθεί. Και αυτό ακριβώς προτείνουμε. Να ανατεθεί δηλαδή στην Κομισιόν η δυνατότητα τροποποίησης μετά από σωστές βέβαια διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες να τροποποιήσει λέω τα παραρτήματα για να μπορέσει να προσαρμόσει τα κατάλαγα. Και βέβαια υπάρχει αυτή η διαδικασία σιωπή ε, του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, δηλαδή να περιμένω τρεις μήνες πριν από την θέση σε ισχύ. Και βέβαια υπάρχει και η κατεπίγουσα διαδικασία που προβλέπεται στην πρόταση. στην περίπτωση κατά την οποία κάτι τελείως καινούριο που δεν έχει στο παρελθόν ληφθεί υπόψη παρουσιαστεί. Στην περίπτωση αυτή προβλέπονται έξι εβδομάδες αν όχι λιγορότερο. για να προσαρμοστούν τα παραδείγματα και να απογορευτεί η εμπορία και η διάθεση. Τελευταίο σημείο είναι βέβαια η ευθύνη των κρατών μελών. Εδώ ισχύει η επικουρικότητα προφανώς και υπάρχει μια μεταβατική περίοδος 36 μηνών που θα ισχύει και για την ε, επεξεργασία των νησιών πάνω από το κατόφλι αυτό, ούτως ώστε να μην εκπληγεί κανένα την ημέρα που θα τεθεί σε ισχύ η οδηγία αυτή και να έχει κάποιους παλιά αποθέματα αυτών των επικίνδυνων ουσιών στο σπίτι του. Είναι λοιπόν σχετικά γενναιόδοροι και πρακτικοί κανόνες, νομίζουμε, και δεν περιμένουμε να υπάρχουν αντιφατικές συζητήσεις. Το Συμβούλιο Αύριο θα αρχίσει στην ε, τεχνική ομάδα εναρμόνισης για την εσωτερική αγορά να εξετάζει το θέμα και ελπίζουμε ότι το Συμβούλιο θα προχωρήσει αρκετά γλυκόρα. Αυτή είναι τουλάχιστον η ιδέα που μας έχουν δώσει. Τόσο ώστε μέχρι τα τέλη του έτους να μπορέσουμε κατά κάποιο τρόπο να υπάρχει συμφωνία μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων. Αυτά από πλευρά μα και πρόεδρε. Σα ευχαριστώ. Thank you. The rapporteur, Mr. Thank uh, Η πρόταση του Κομισιόν είναι σαφή. Είναι διαφορετική κατάσταση στα κράτη-μέλη και στα 27 δεν το επιθυμούμε αυτό. Υπάρχουν κάποιε ουσίε που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τρομοκράτε και νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε αυστηρές, αυστηροί να πούμε ότι ε, δεν είναι διαθέσιμα τόσο εύκολα πια τα επικίνδυνα υλικά κάποιες ανησυχίες που υπάρχουν ε, είναι ο κατάλογος. Είναι πλήρως ο κατάλογος. Ήδη έχω κάνει κάποιες συζητήσεις με την βιομηχανία. Ε, νομίζω ότι θα πρέπει να προσταθούν και άλλα στον κατάλογο και αυτό θα ήταν καλό. Αλλά πρέπει να προσέξουμε ότι σε περίπτωση που δώσουμε άδειε σε κάποιου ανθρώπου για να πολλούν τέτοιο υλικό σε άλλε συγκεντρώσει από το φυσιολογικό, αν ε, δούνε περίεργε συναλλαγέ, τότε θα πρέπει να τις αναφέρουν απευθείας στις δικαστικές αρχές. Ε, βεβαίως ε, υπάρχει και θέμα προστασίας δεδομένων το οποίο θα πρέπει να εξασφαλίσουμε και η Επιτικομισία θα πρέπει να το δει αυτό. Κατά τα λοιπά, φαίνεται ότι είναι μια πρόταση την οποία μπορώ να στηρίξω και νομίζω ότι θα πρέπει να τη διεκπαιρεώσουμε το συντομότερο δυνατόν. Ευχαριστώ. Thank you, Mr. Εγώ ευχαριστώ κύριε Μούλτερ που ήσασταν τόσο συνεκτικός. Η κυρία Ματιό είναι η σκιώδη συγκεντρία. Ευχαριστώ πρόεδρε. Έχω την ίδια αντιμετώπιση με του κυρίου Μιλντερ. Η Europol μας είπε ότι ορισμένες τρομοκρατικές επιθέσεις έγιναν με χρήση προϊόντων που βρίσκουμε στο εμπόριο, δηλαδή εραστεχνικές βόμβες και θα πρέπει να δούμε, να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα. Νομίζω, όπως είπε και ο εισηγητής, ο κατάλογος των παραρτημάτων είναι και το ζωτικότερο ζήτημα, Άρα ίσως θα πρέπει να ολοκληρώσουμε με τα παραρτήματα, τα παραρτήματα και το σύστημα αδειοδότησης είναι κάτι το περίπλοκο ίσως. Ίσως θα μπορούσαμε να βρούμε κάτι πιο απλό και λιγότερο γραφειοκρατικό και λιγότερο δαπανηρό για τα κράτη-μέλη, για την καταπολέμηση της ε, τρομοκρατίας έτσι ώστε να προωθήσουμε την ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα έχουμε την ευκαιρία να θίξουμε αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ. Αν δεν υπάρχουν άλλα σχόλια, από... ναι, έχετε το λόγο. Ο κύριος Μπρόνς. Δεν είμαι ενθουσιώδης ως προς την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία ως όπως είναι γνωστό. Κάτι όμως με απασχολεί και είναι το εξής, ότι αυτή η νομοθεσία θα τεθεί σε ισχύ σε 36 μήνες. Στο μεταξύ, θα καλέσουμε τη βιομηχανία και το λιανικό εμπόριο να έχει μία άτυπη, ένα άτυπο μήτρο αγορών κάτι τέτοιο θα προανακοινωθεί και φαντάζομαι ότι αυτοί που θέλουν να σωρεύσουν αυτές τις πληροφορίες θα το προωθήσουν το θέμα. Υπάρχει κάποιος μηχανισμός έτσι ώστε τουλάχιστον να έχουμε ένα μητρό αυτών που αγοράζουν αυτές τις ουσίες για να μην τις αποθηκεύσουν εκ των προτέρων. Κάποιος έλεγχος τέλος πάντων. Γιατί αν θέλω εγώ να αγοράσω μια χιουσία από το φαρμακείο, τότε, από όσο ξέρω τώρα δεν υπάρχει κανένας περιορισμός και κανένας δεν γνωρίζει την ταυτότητά μου. Και αυτό με απασχολεί όλος ιδιαιτέρως. Thank you. Εάν δεν Υπάρχουν άλλα σχόλια. Ο κύριο Σίφερ κάτι θέλει να μας πει. Uh, Ευχαριστώ. Όπως είπα στην πρώτη μου παρέμβαση, ήρθαμε σε επαφή με τη βιομηχανία από τη Μόνιμη Επιτροπή Πρόδρομων Ουσιών για το νέο πρόγραμμα δράσης για τις εκρηκτικές ύλες και αυτή η Επιτροπή συνεδριάζει όσο βρισκόμαστε εμείς εδώ. Ήρθα σε επαφή με τις αρχές ασφαλείας και τις ε, συναφείς επιχειρήσεις που ασχολούνται με τις πρόδρομες ουσίες και τις εκρηκτικές ύλες. Θα σας πληροφορήσουμε για την εξέλιξη των διαβουλεύσεων και Γνωρίζουμε τι έχει προταθεί, πώς έχει το χρονοδιάγραμμα, καθώς και όλες τις ουσίες που έχουν καταμετρηθεί. Και γνωρίζουμε, γνωρίζει ο καθένας τι χρησιμοποιεί στο εμπόριό του ή στο εμπόριο με άλλους και έχουν ε, ε, σε θελούσια βάση αρχίσει αλλαγές ως προς την παραγωγή, δεν υπάρχει υποχρέωση και όλα αυτά αποτελούν εκούσια, μια εκούσια επιλογή. Εάν βεβαίως τεθεί σε ισχύ το όλο πλαίσιο μέχρι το τέλος του έτου τους, τότε ακόμα και αυτοί που θα έχουν προσχωρήσει αργά θα πρέπει να αρκεστούν σε αυτό το πλαίσιο. Αν δεν υπάρχουν άλλα σχόλια, τελειώνουμε για σήμερα. Σας υπενθυμίζω ότι θα έχουμε την υποβολή της έκθεσης 16-17 Μαρτίου. of the Libe Όταν συνεδριάσουμε ως Επιτροπή. Αυτά για σήμερα. Αύριο θα αρχίσουμε στις 9. Σας ευχαριστώ. Γεια σας.